Verehrte Kolleginnen und ο κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω την συνεδρίαση και την ακρόαση. Σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό και βεβαίως όλος ιδιαιτέρως τον υποψήφιο Επίτροπο για θέματα υγείας, τον δόκτορα Τόνιο Μπόργκ και θα εξηγήσω με λίγα λόγια την διαδικασία, ώστε όλοι να γνωρίζετε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε στη διάθεσή μας τρεις ώρες. Πρώτα θα λάβει το λόγο ο ίδιος ο Δόκτωρ Μπόρκ για να κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση 10 λεπτών. Μετά θα έχουμε στη διάθεσή μας 155 λεπτά για να θέσουμε ερωτήσεις. Αυτός ο γύρος ερωτήσεων έχει κατανεμηθεί ως εξής. θα τεθούν 10 κάπως μακροσκελέστερες και 15 ε, σύντομες ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής και στο ε, μεταξύ θα τεθούν από την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών 7 μακρές και 3 σύντομες ερωτήσεις, καθώς και δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής αυτής, κ. Χάρμπορ, τον οποίο καλωσορίζω επίσης στην παρουσά ακρόαση. Η δε τρίτη συμμετέχουσα επιτροπή είναι η Επιτροπή Γεωργίας, που θα έχει τη δυνατότητα να θέσει πέντε σύντομες ερωτήσεις. Οι μακρέ ερωτήσει θα είναι κάπως σαν πινκ-πονγκ. Ένα λεπτό για την αρχική ερώτηση, δύο λεπτά για απάντηση από πλευρά του υποψηφίου και μετά θα διατεθούν ακόμη 45 δευτερόλεπτα για τον ερωτώντα εφόσον θέλει να υποβάλει ε, δεύτερη ερώτηση. Οι δε σύντομες ερωτήσεις θα είναι 3 λεπτά και 50 δεύτερα για την ερώτηση και 2 λεπτά για την απάντηση. Και δικό μου καθήκον και καθήκον του κ. Χάρμπορ είναι σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα της Ευγένειας να φροντίσουμε ώστε να διεξαχθεί η συζήτηση αυτή σε ευγενή και ομαλή ατμόσφαιρα. Θα φροντίσουμε λοιπόν ώστε να είναι δικαία η ακρόαση του υποψηφίου. Για εμάς, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και για όλες και όλους τους υπολείπους, σήμαινε η αλλαγή αυτή, ήταν μια απότομη αλλαγή και από αυτού επιθυμώ να δηλώσω ότι η αλλαγή αυτή στο πρόσωπο του Επιτρόπου θα πρέπει να διαχωριστεί από την σημερινή ακρόαση και να, έχουμε, να δώσουμε σε αυτούς σήμερα την ευκαιρία να υποβάλουμε ερωτήσεις και να λάβουμε ε, απαντήσεις που να μας διαφωτίσουν. Θα αρχίσουμε λοιπόν τώρα και θα ήθελα πρώτα να δώσω στον υποψήφιο Υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας, κύριο Μπόρκ, την δυνατότητα να λάβει το λόγο για 10 λεπτά και να κάνει έτσι την πρώτη του εισαγωγική τοποθέτηση. Θα παρακαλέσω τώρα πάλι όλες και όλους, επιμένει ο πρόεδρος, όλες και όλους, είπα προηγουμένως ότι πρόκειται σήμερα είναι η ημέρα της ευγενία. Και αυτό επιβάλλει σε όλες και σε όλους να καθίσουν, να αναζητήσουν την θέση τους, να καθίσουν, να υπάρξει ησυχία στην αίθουσα έτσι ώστε ο δόκτωρ Μπόρκ να μπορέσει να προβεί στην εναρκτήρια δήλωσή του. Έχετε το λόγο, δόκτωρ Μπόρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε αυτό το κτίριο, σε αυτό το θεσμικό όργανο προκειμένου να ανταλλάξω απόψεις με τους ευρωβουλευτές ως υποψήφιος επίτροπος που εφόσον οριστώ θα είμαι υπεύθυνο για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών. Το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι για μένα αυτό που ονομάζω η Ευρώπη σε πρώτο επίπεδο. Η βάση αυτό που επίσης λέω το χαρτοφυλάκιο των ανθρώπων διότι καλύπτει θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των ασθενών και των καταναλωτών. Ήμουνα βουλευτή τα τελευταία 20 χρόνια και μέλος της κυβέρνησης στη Μάλτα για τα τελευταία 14 χρόνια, έχοντα καλύψει διάφορα χαρτοφυλάκια, μεταξύ άλλων και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Εφόσον οριστώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου αυτή προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω την σχέση μου μαζί σας να την κάνω μια σχέση πλήρους συνεργασίας. Και όχι μόνο επειδή το Κοινοβούλιο έχει αποφασιστικό ρόλο στην νομοθεσία, αλλά γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό που πρέπει να κάνω. Θα φροντίσω η αυτή να μην είναι ανοιχτή, χωρίς εμπόδια και να είμαι ειλικρινής και τιμίος μαζί σας. Δεν σας υπόσχομαι το κατόρθωτο, αλλά σκοπεύω να δουλέψω προκειμένου να πετύχω όσο γίνεται περισσότερα μαζί σας. Θέμα ανεξάρτητος, θα είμαι αντικειμενικός, αλλά πάνω απ' όλα θα είμαι Ευρωπαίος. Έχω αφοσιώσει το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής μου ζωής, τα τελευταία δηλαδή 30 χρόνια, προκειμένου η Μάλτα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί? Γιατί πιστεύω στις ευρωπαϊκές αξίες. Και είναι τιμή για μένα που πέτυχα τη στήριξη των δύο μονοπολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο της Μάλτας, κάτι το οποίο πρέπει να σας πω όσον αφορά την παράδοση της χώρας μου, είναι μια μεγάλη πρόκληση και μεγάλη επιτυχία από μόνο του. Για το υπόλοιπο της εντολής μου θα φροντίσω να προσφέρω στους ασθενείς και τους καταναλωτές αυτό που εγώ ονομάζω στα αγγλικά 3C, τα 3C, Continuity, confidence και commitment, δηλαδή να διασφαλίσω τη συνέχεια, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και να φροντίσω επίσης να φέρω σε πέρα στις δεσμεύσεις μου. Όντως δεσμεύομαι πλήρως από τις υποχρώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέχρι τώρα. Θα φροντίσω για πρωτοβουλίες όσον αφορά την αναλλακτική επίλυση διαφορών, την ε, online επίλυση διαφορών, πράγματα τα οποία ήδη βρίσκονται στο αυλάκι, όπως επίσης οι κλινικές δοκιμές, θέματα που έχουν να κάνουν με τα ιατρικά μηχανήματα κτλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι η πολιτική προς όφελος του καταναλωτή μπορεί να πετύχει και την εμπιστοσύνη υπέρ της εσωτερικής αγοράς, αλλά μπορούμε να πετύχουμε και εμπιστοσύνη των καταναλωτών βάσει δοκιμών που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Αυτό τι σημαίνει πιο συγκεκριμένα. Στον τομέα της υγείας, η παριθμόν ένα προτεραιότητά μου είναι πολύ γρήγορα να παρουσιάσω μια φιλόδοξη πρόταση όσον αφορά τα προϊόντα καπνού. Γιατί το κάπνισμα είναι η κυριότερη αιτία πρώιμων θανάτων. 95% όλων των καπνιστών αρχίζουν να καπνίζουν πριν φτάσουν στα 25 χρόνια ηλικία. Και το 70% αρχίζει να καπνίζει μάλιστα πριν και από τα 18. Ήμουν 16 όταν κάπνισα το πρώτο μου τσιγάρο. Θα φροντίσω λοιπόν για μια φιλόδοξη πρόταση η οποία θα αναθεωρήσει την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Μια πρόταση η οποία θα προσφέρει μια καλή λειτουργία στην εσωτερική αγορά με υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Θα είναι μια πρόταση η οποία θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Διαθέτουμε τα εργαλεία. Ελπίζω ότι θα μπορώ να βασιστώ σε εσά για να ολοκληρώσω το έργο μου. Δεύτερη προτεραιότητά μου είναι η βελτίωση τη κατάσταση όσον αφορά του ασθενεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντα τα κράτη-μέλη στι δικέ του προσπάθειε για να προσαρμοστούν στι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε εξαιτία ε, των ε, χρόνιων ασθενών που αυξάνουν όλο και περισσότερο και τη γύρανση του πληθυσμού, παρά τι οικονομικέ ε, δυσκολίε και περιορισμού. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, διασφαλίζει για όλους το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία. Θα φροντίσω λοιπόν να χρησιμοποιήσω ό,τι μέσα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και θα σεβαστώ απόλυτα την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών σε αυτό το τομέα. Είμαι πεπισμένος όμως ότι μαζί έχουμε πολλά να κερδίσουμε μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον και βάζοντας μαζί τους πόρους μας. Γιατί η υγεία είναι μια επένδυση. Δεν είναι μόνο μία δαπάνη και, απόλα, όλα, και πάνω απ' όλα αποτελεί αυτή καθεαυτή αυτή μία αξία. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου τώρα να συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα, που είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά λοιπόν την πολιτική καταναλωτών, θέλω να σας υποσχεθώ ότι εφόσον επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου στη θέση του Επιτρόπου, πρόθεσή μου είναι να προστατεύσω τα συμφέροντα των καταναλωτών και να είμαι ένας πρωταθλητής όσον αφορά τα θέματα καταναλωτών. Αρχή μου είναι να διασφαλίσω ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο έτσι ώστε τα δικαιώματα των καταναλωτών να γίνει πραγματικότητα, κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την ενιαία αγορά βέβαια, η οποία πρέπει να προσφέρει ωφέλη προς τους καταναλωτές. Η ενιαία αγορά αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Πρέπει να ενισχύσουμε επίσης την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά και έτσι πιστεύω θα βοηθηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρει το δρόμο της ανάκαμψης. Ένα βασικό θέμα που απασχολεί του καταναλωτέ είναι η ασφάλεια. Στις αρχές επόμενη χρονιά θα υποβάλω μαζί με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη ένα πακέτο όσον αφορά την ε, ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει να απλοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες κανόνες και να βελτιωθεί η εποπτεία της αγοράς και να τηρούνται οι κανόνες. Το πακέτο αυτό θα αποτελέσει την έκφραση του γεγονότος ότι η ασφάλεια δεν ε, πρέπει να είναι κάτι που βλέπουμε σαν αντιπαράθεση με την ε, ανταγωνιστικότητα. Αντίθετα, πρόκειται για μια επένδυση που κάνουμε στην ανταγωνιστικότητα, γιατί έτσι το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά μεγαλύτερη αξία. Ε, μια άλλη πρωτοβουλία κλειδί, νομοθετική πρωτοβουλία, που θα υποβάλω στις αρχές της επόμενης χρονιάς, εφόσον αναλάβω το χατοφυλάκιό μου αυτό, μαζί με τον Επίτροπο Μπαρνιέ, θα είναι μια πρωτοβουλία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και αυτό προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πληροφορίες με διαφάνεια και ότι θα μπορούν να διαχειριστούν τους λογαριασμούς τους όπως θέλουν. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, στον τομέα των τροφίμων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει πολλά. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο που βασίζεται στις υψηλές προδιαγραφές, στις επιστημονικές που έχουμε. Και όντω η επιστήμη θα με καθοδηγεί όταν θα πρέπει να παίρνω δύσκολες αποφάσεις. Γιατί το βασικό είναι να εφαρμόζουμε ορθά τους κανόνες που ήδη υπάρχουν. Πάντα μπορούν να βελτιωθούν. Θα είμαι πρόθυμος να προτείνω πακέτο προτάσεων όσον αφορά τα φυτά, ε, τα ζώα, την προστασία των ζώων, τους σπόρους, όπως επίσης τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και τις δαπάνες που κάνουμε για όλα αυτά για την περίοδο 2014 με 2020. Και βέβαια θα δώσω ιδιαίτερη σημασία στους ελέγχους. Και βέβαια Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την κλωνοποίηση, να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Δικιά μου φιλοδοξία είναι να υποβάλω μια νομοθετική πρόταση επίση και για τα νέα τρόφιμα την επόμενη χρονιά. Τώρα, για να έρθω στην προστασία των ζώων. Η προστασία των ζώων είναι ένα σημαντικό θέμα, μια βασική ευρωπαϊκή αξία, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Εξάλλου, οι ίδιες οι συνθήκες αναφέρονται στα ζώα σαν ε, όντα. Γι' αυτό θα επικεντρωθώ στο να βελτιώσω την ε, ζωή των ζών εφαρμόζοντας ακόμα καλύτερα τους ήδη υπάρχοντες νόμους. Διάφορες δράσεις που έχουν γίνει και προσφυγές εναντίον ε, χωρών μελών έχουν ήδη αποφέρει καρπούς και όσον αφορά τις οτόκες ε, όρνηθες και θα φροντίσω επίσης να συνεχίσω την ίδια προσέγγιση προκειμένου να διασφαλίσω την εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων κανόντων και στον τομέα της μεταφοράς των ζώων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σε καιρούς οικονομικής κρίσης υπάρχει η τάση να μειώνουμε τις δαπάνες. Για μένα, ο σημαντικός παράγοντας είναι να διασφαλίσω ότι όταν υπάρχει περικοπή στις δαπάνες, η περικοπή αυτή να γίνεται με φύ τρόπο και να συνειδητοποιούμε πάντα ότι πρέπει να προστατεύουμε τους αδύναμους και τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας. Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει ποτέ την κοινωνική της πηξίδα. Η υγεία και οι πολιτικές για τον καταναλωτή είναι τομείς όπου δράσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι από το οποίο εποφελούνται οι καταναλωτές και οι ασθενείς. Εάν κερδίσω την εμπιστοσύνη σας, σας υπόσχομαι ότι θα υπηρετήσω με όσο γίνεται μεγαλύτερη και περισσότερη ενέργεια. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα χρησιμοποιήσω όλες τις δεξιότητές μου ώστε να πετύχω στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους και τις πολιτικές για μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ ο πρόεδρος κ. Γκρότε. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Μπόρκ. Θα αρχίσει τώρα ο γύρος των ερωτήσεων από πλευρά συντονιστών. Για μια σύντομη ερώτηση, ο κύριος Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ. Δεν έχει μικρόφωνο ο κ. Λίζε. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του κύριου Λίζε. Τώρα λειτουργεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε υποψήφιε Επίτροπε για τα εισαγωγικά σας λόγια. Επιτρέψτε μου να επανέλθω με μια ερώτηση για την οδηγία για τον καπνό. Η πρόταση αυτή είχε αναβληθεί κατ' επανάληψη στο εσωτερικό της Κομισιόν και ορισμένοι πιστεύουν, αντίθετα με αυτά που ανακοινώσατε, ότι ενδέχεται η πρόταση αυτή να είναι και νεκρή. Η πλειοψηφία από εμά εδώ θα ήθελε πράγματι να υποβάλλετε τη σχετική πρόταση σύντομα. Ερώτηση. Έχετε χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να μας πείτε λεπτομέρειες. Έχετε και κάποιες ουσιώδεις λεπτομέρειες που θα θέλατε να δείτε στην πρόταση αυτή. Και εάν διαθέσετε όλη την ενέργειά σας, θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει καμία πλέον καθυστέρηση. Ο Δόκτωρ Μπόρκ για δύο λεπτά. Πιστεύω ότι η οδηγία για τον καπνό δεν είναι νεκρή. Είναι ζωντανή και σπαρταρά. Στην πολιτική μου σταδιοδρομία σπανίως υπεσχέθην πράγματα εκτός από αυτά που μπορώ να εκπληρώσω διότι αυτή τη στιγμή υποσχεθεί κανείς κάτι μπορεί να του έρθει πάλι ως μπούμεραγκ. Αυτό που μπορώ να σε υποσχεθώ είναι το εξή. Εάν τελικώς εγκρίνεται τον διορισμό μου η πρώτη μου ενέργεια θα είναι να στείλω την οδηγία για τον καπνό στις υπηρεσίες για διαβούλευση και να προωθήσω την έγκριση της οδηγίας. Δεν εφευρίσκω κανένα χρονοδιάγραμμα, τα έχω εξετάσει και οφείλω να πω ότι προς την κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνθηκα από τον ίδιο τον πρόεδρο κ. Μπαρόσο. Αυτά που σας λέω λοιπόν εδώ είναι πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι σημαντικό επίσης, εάν συμβεί αυτό και βέβαια θα συμβεί, είναι σημαντικό εσείς να με υποστηρίξετε έτσι ώστε να υλοποιηθεί η οδηγία αυτή στη διάρκεια της παρούσης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, η οδηγία βρίσκεται ακόμα στην εμπιστευτική φάση της διαδικασίας, διότι ακόμη δεν έχει εγκριθεί από το συλλογικό όργανο των επιτρόπων. Μπορώ όμως να σας πω με λίγα λόγια προσωπικές μου απόψεις για το περιεχόμενό της. Πρώτα πιστεύω ότι τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να έχουν και την πορφή προϊόντων καπνού και θα πρέπει να έχουν και τη γεύση των προϊόντων καπνού. Η οδηγία αυτή βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης, η οποία διασφαλίζει στην ενιαία αγορά υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Και γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους όλες οι στατιστικές δείχνουν ότι υψηλό ποσοστό εκείνων που καπνίζουν για πρώτη φορά το κάνουν πραγματικά σε πολύ νεαρή ηλικία. Και υπάρχουν και κάποιες τάσεις. Οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο από τους άνδρες, για παράδειγμα. Άρα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, όχι μόνο, με συγχωρείτε, όχι μόνο με το να εμφανίζονται, να έχουν την εμφάνιση προϊόντων καπνού, αλλά και πραγματικά το ίδιο και στις διαφημιστικές τους εκστρατείες. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πράγματα που θα πρέπει να περιληφθούν. Για παράδειγμα, να μην γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ διαφόρων προϊόντων καπνού. Η επόμενη ερώτηση από την κυρία Μακάβαν. Είμαι από αυτή την πλευρά εδώ, κύριε Επίτροπε. Μιλήσατε για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και ιδίω για τον χάρτη των ανθρώπινων, των θεμελιδών δικαιωμάτων. Πώς όμως συμβιβάζονται αυτά με ορισμένα πράγματα που ακούμε για τις δραστηριότητές σας στην Μάλτα και κυρίως για δικαιώματα γυναικών και την άμβλωση, όπου όχι μόνο φροντίσατε να γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία στην Μάλτα, καθιστώντας παράνομη συνταγματικά την άμβλωση, αλλά έχετε περιορίσει και τις μετακινήσεις γυναικών που ενδέχεται να μεταβούν στο εξωτερικό για να προβούν σε άμβλωση. Δεύτερο, για θέματα μη διακρίσεων ε, των προσώπων σχετικά με τον ε, ερωτικό τους προσανατολισμό. Έχουμε ακούσει ότι έχετε ζητήσει να μην εφαρμόζεται πλήρως ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την ελεύθερη διακίνηση και ότι στην συζήτηση για τα ίσια δικαιώματα έχετε ζητήσει να προστατεύονται μόνο εκείνοι οι οποίοι αξίζουν την προστασία. Πώς συμβιβάζονται οι δηλώσεις αυτές με κάποιον που θέλει να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, παρακαλώ να σέβεστε τα χρονικά όρια. Οπωσδήποτε, Πρόεδρε, για το θέμα των αμβλώσεων. Η συνθήκη είναι πολύ σαφής για το θέμα αυτό. Είναι πολύ αρμοδιότητα των 100 μελών το αν θα επιτρέψουν ή όχι κάτι τέτοιο. Ως Ευρωπαίος λοιπόν Επίτροπος θα συμμορφωθώ με τις συνθήκες και με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα σεβαστώ επίσης την αρχή της επικουρικότητας. Δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της αρχής αυτής να εμπλέκεται στην άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι, διότι έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα σε εφημερίδα που αναφέρει ότι πριν από 14 χρόνια, όταν τέθηκε το ζήτημα αν πρέπει να επιτραπεί σε μία Μαλτέζα πολίτη που ήθελε να, να υποβληθεί σε άμβλωση στη Μεγάλη Βρετανία, αν θα της επιτραπεί λοιπόν αυτό ή όχι, από το 1998 τότε τέθηκε το θέμα εάν θεωρείται νομικός ε, ορθό ή όχι να μεταβεί εκτός Μάλτας ε, για το σκοπό αυτό ή όχι. Και εγώ δήλωσα τότε ότι ενώ έχω δηλώσει προσωπικά ότι είμαι κατά των αμβλώσεων, θεωρώ ότι από νομικής άποψη, η γυναίκα αυτή που μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έκανε τίποτε το παράνομο. Το ποινικό δίκαιο στη Μάλτα περιορίζεται στην άσκηση του δικαίου εντό τη χώρα. Επίσης υπήρξε και άλλη μια δήλωση που έλεγε ότι αντιδρώντας στα σχόλια του κυρίου Μπόρκ, ο κύριο Τάδε είπε ότι το βρήκε κάπω παράξενο ο Δόκτωρ Μπόργκ, μέλος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, να λέει ότι η κυρία αυτή δεν έκανε τίποτε το παράνομο. Τώρα, για το σεξουαλικό προσανατολισμό. Φέτος ε, ασχοληθήκαμε με, την, με νομοσχέδιο για την ε, ρύθμιση των σχέσεων εκτός γάμου, ιδίως των σχέσεων του ιδίου, στο, του ιδίου φύλου, καθώς και την τιμωρία για πράξεις άσκησης βίας λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού. Στη χάρτα αυτό απηχείται στο σημείο 21 και βεβαίως στη Μάλτα γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα, χάρη και στη δική μου παρέμβαση. Κυρία Μακάβαν. Και πώς αυτά θα έχουν επιπτώσεις ε, στις αποφάσεις του Κολεγίου των Επιτρόπων, λόγω χάρη για τα βλαστοκύτταρα ή για τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα δικαιώματα σεξουαλικής αναπαραγωγής των δικαιών σε άλλες χώρες. I shall abide by all the Όσα προγράμματα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα σεβαστώ πλήρω και να εξηγήσω γιατί. Τα προγράμματα αυτά έχουν ήδη εγκριθεί Υπάρχει η αρχή της ε, ομαδικότητας και διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές νομοθεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθείτε η θέση που ισχύει και θα πρέπει να προστατεύετε στην κάθε χώρα όπως ορίζει η συνθήκη. Άλλο οι προσωπικές μου πεπιθήσεις. Οι διάφοροι νόμοι έχουν εγκριθεί βάσει των νομοθεσιών των κρατών μελών και για τι χώρε που είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτές που βρίσκονται εκτός. Κατά τα άλλα θα παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητα. Τι σημαίνει η αρχή αυτή, ότι κάθε χώρα είτε επιτρέπει την άμβλωση ή όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει και δεν μπορεί κανείς να παρέμβει στις αποφάσεις της χώρας αυτής άσχετα εάν αυτέ συμφωνούν με τι προσωπικέ μου πεπιθήσει. Διότι θα είμαι πάνω απ' όλα επίτροπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα είμαι Μαλτέζο επίτροπε, Θα είμαι Ευρωπαϊκό επίτροπο που έχει διοριστεί από τη χώρα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στέβης. Κύριε Επιτροπέ, δεν αμφισβητώ τι ικανότητέ σα, αλλά τι απόψει σα. Μπορεί να είναι σχετικό συντηρητική χώρα η Μάλτα, αλλά ακόμα και με τα πιο συντηρητικά πρότυπα, εσεί φαίνεται να είσαστε αρκετά ακραίο. Έχετε ένα ιστορικό ότι έχετε κάνει κάποιε ομοφοβικέ παρατηρήσει για τα ζευγάρια ομοφυλοφίλων. Έχετε φέρει αντιρρήσει για το νόμο διαζυγίου τη Μάλτα και έχετε προσπαθήσει να, τα, να παρεμποδίσετε την πρόοδό του και επίση το ίδιο με τη δωρεά οαρίων και σπέρματο. Εδώ, στην ακρόαση αυτή, έχουμε ακούσει και μέχρι εδώ τις απόψεις ε, υποψηφίων σε προκλογικέ εκστρατείες ως τώρα, καθώς και στην όλη διαδικασία υποψηφίων. Γιατί εδώ λοιπόν να σας εγκρίνω, όταν υπήρξατε υπουργό και εκφράσατε τόσο συντηρητικές απόψεις. Η επιλογή είναι ελεύθερη. Εδώ καλείστε να δείτε κατά πόσον τοποθετούμε σαφώς ως προς όσα λέω. Ουδέποτε υπήρξα εκτός, κατά των σχέσεων εκτός γάμου, όποιος σεξουαλισμό, τουλισμου και αν είναι, ενέκρινα μια σειρά από νόμους ώστε να ρυθμιστούν οι εκτός γάμου σχέσεις, είτε είναι ετεροφιλοφιλικές είτε ομοφιλοφιλικές, και βεβαίως ο νόμος αυτός είναι καλύτερος από αυτόν που υπάρχει, που, από την απουσία νόμου σε πολλά κράτη-μέλη. Εφόσον ο νόμος αυτός εγκριθεί, σημαίνει ότι θα υπάρξουν νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και μια σχέση συμβίωσης θα μπορεί να καταγραφεί ε, και να επιτραπεί στα ζευγάρια του ίδιου φίλου ή διαφορετικών φίλων να ζουν μαζί. Αυτό για μένα είναι ένα βήμα πρόοδου. Και θα σημαίνει ότι θα μπορεί να δημιουργείται οικογένεια και με την παρουσία νομίμων συντρόφων. Δεν τοποθετήθηκα λοιπόν κατά των σχέσεων ε, και των ζευγών ιδίου φίλου, απλώς ότι θα ήταν ε, άδικο για, τους γάμους, για τις νόμους εκμεστώσεων στη Μάλτα να ορίζει τις σχέσεις εκτός γάμου χωρίς να υπάρχει ένας νόμος για αυτό καθε το θέμα. Δεν μπορεί να επιβάλλεται κάτι ε, εμέσως πλην σαφώς σε έναν σπιτονικοκύρη από την κυβέρνηση. Στον νέο νόμο αυτό θα διευθετείται και, τους, ε, και για τις εκμισθώσεις που θα ξεκινάνε από ένα χρονικό σημείο και μετά. Αυτή ήταν η μόνη παρατήρηση που έκανα και ουδέποτε έκανα επικριτικές παρατηρήσεις για το αν θα πρέπει να ανοιχτούμε τους ομοφυλόφιλου ή όχι. Ουδέποτε είπα κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να διαβάσετε ακριβώς την καταγραφή των σχολείων μου για να δείτε τι επικριτικά σχόλια ανέφερα. Ίσα ίσα για την καταπίεση των ανθρώπων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, εγώ ένεκρινα νόμους που καταπολεμούν τα φαινόμενα αυτά. Ευχαριστώ για αυτή την απάντηση. Αλλά υπάρχουν ε, αντιφατικές τελικά μαρτυρίες για το τι σχόλια κάνατε. Και εδώ μπορώ να θυμίσω και το Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Όπου η κλασική προσέγγιση ήταν αν δεν ξέρετε ψηφίστε όχι. Όμω, ό,τι αφορά το δικό σα χαρτοφυλάκιο, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι προσωπικέ σα πεπιθήσει για τα κοινωνικά θέματα δεν θα επηρεάσουν και το πώ θα εγκρίνετε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα ασκήσετε διακριτική μεταχείριση. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα βασιστώ και θα βασίσω την πορεία μου στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτή η χάρτα μας απασχόλησε και στο Υπουργείο μου για το κατά πόσον θα πρέπει να την κυρώσει η Μάλτα ή όχι. Ήμουν υπέρ της κυρωσής της. Νομοθεσία για την κατάργηση της θενατικής ποινή. Είναι κάτι που το υποστήριξα. Επίσης υποστήριξα νομοθεσία για την ε, ε, νομιμοποίηση των τέκνων που γεννούνται εκτός γάμου. Επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί μια εικοσαετία. Έχω δώσει διαλέξει στο Πανεπιστήμιο για το θέμα αυτό. Είναι δικό μου θέμα. Είναι κάτι που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ ω θέμα αυτό. Και είναι σαφέ το άρθρο 21 ότι οποιαδήποτε διακριτική συμπεριφορά, όχι μόνο βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού ή βάσει του φύλου, ή είναι κάτι που απαγορεύεται και βεβαίω θα το σεβαστώ. Αυτό με αυτό ω βάση θα χαράξω πορεία. Τη χάρτα των θεμελιδών δικαιωμάτων. Thank you Κυρία Χάση. Ευχαριστώ. Θέλω να συνεχίσω μετά από αυτά που είπαν ε, η κυρία Μακάβεν και ο κύριος Ντέιβις. Είναι σημαντικό το ότι την εποχή που ήσασταν υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας, η Μάλτα ήταν η χώρα η οποία μπόδισε στήριξη για σημαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι η πλατφόρμα του Καΐρου. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσο εσείς θα υποστηρίζατε την σημασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών ε, δικαιωμάτων συνολικά. Θα ήθελα να έχω τις απόψεις σας για τα θέματα αυτά για παράδειγμα για την καταπολέμηση του AIDS, της επιδημίας αυτής και γενικότερα για την προστασία της υγείας των ε, πολιτών γενικότερα. Απάντηση. Ήμουν υπουργό εξωτερικών τέσσερα χρόνια και ποτέ δεν ασχολήθηκα με θέματα ανάπτυξης. Οπότε πρέπει να ρωτήσετε τον αρμόδιο υπουργό γι' αυτό, αλλά εντάξει, πολλά χαρτοφυλάκια ασχολούνται με την ε, ανάπτυξη, είναι αλήθεια. Εγώ είπα ότι θα συμμορφωθώ με τις αποφάσεις που θα ληφθούν βάσει της αρχής και της επικουρικότητας. Όσον αφορά το AIDS και άλλες ασθένειες, ευτυχώς σήμερα δεν είναι η ίδια μάστιγα όπως ήταν κατά το παρελθόν. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας όσον αφορά την καταπολέμηση του AIDS. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη, στην διάγνωση και στη θεραπεία. Και ιδιαίτερα να απαλληφθεί ο στιγματισμός των ατόμων εκείνων που υποφέρουν από αυτή την τραγωδία των μοντέρνων καιρών. θα πάω και στην διάσκεψη που οργανώνει ο ΙΕ όσον αφορά το AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί πράγματι είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ε, διαβεβαίω λοιπόν κυρία Χάση ότι εφόσον είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος θα φροντίσω γι' αυτό. Καλώς, ευχαριστούμε. Η το Χάση να συμπληρώσει. Θα ήθελα να διευκρινίσω λίγο το θέμα. Ε, συμφωνείτε μαζί μου και με την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ότι σεβόμενοι την, ε, τους ομοφιλόφιλους η εκπαίδευση των εφήβων όσον αφορά θέματα σεξουαλικότητας, ε, επιλογών, αναπαραγωγικότητας θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και το θέμα του AIDS και την προστασία της υγείας γενικά. Κύριε Ναι, κύριε Χάση. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα φύλακες διακρίσεων σε όλες τις χώρες μέλη που πρέπει να καταπολεμηθούν και πρέπει να τους εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα και να τους ε, καταστρέψουμε. Άλλες φορές που έχω συζητήσει λέγανε ότι άμα ρωτάει κανείς τι πρέπει να ρωτάει, πρέπει να ρωτάει αν είσαι γκέι ή αν δεν είσαι ή πρέπει να ρωτάει ποιος είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός γενικά. Έχει σημασία η διατύπωση και για τους ανθρώπους αυτούς είναι σημαντικό. Πρόκειται τελικά για μια διάκριση που είναι παρούσα ακόμα σε πολλές χώρες μέλη. Ευχαριστούμε. Μαρίνα για ένα κουδάκι τώρα. Τώρα είναι η σειρά σας. Ευχαριστώ. Την ακρόαση αυτή τη βλέπει η ομάδα μου σαν ευκαιρία αξιολόγηση των γνώσεών σας στο χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβετε. Οι εθνικέ πολιτικές και οι διατάξει για την υγεία είναι τομεί που είναι αρμοδιότητα καθαρά των χωρών μελών. Οι κλινικέ δοκιμές, υπάρχει μια σχετική οδηγία που επικρίνουν διάφορες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τους ευγενείς στόχους, είναι αλήθεια ότι έχει περάσει πάρα πολύς ε, χρόνος και ότι η γραφειοκρατία επιδεινώνεται. Εσείς πώς βλέπετε την πρόταση για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να λεφθούν υπόψη οι ανησυχίες αυτές και πώς εσείς θα δώσετε όθηση σε νέους ε, τομείς. Όσον αφορά την οδηγία για τις κλινικές δοκιμές που συζητιέται αυτή την εποχή. Προτείνεται ακριβώς για τους λόγους που είπατε. Επειδή η υπάρξη μείωση των κλινικών δοκιμών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να παρέμβει με τέτοια οδηγία, όχι για να είναι λιγότερο ασφαλείς οι δοκιμές αυτές, όχι αντίθετα, για να μειωθεί η γραφειοκρατία και για να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες ε, κλινικές δοκιμές, βέβαια μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας. Και πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των ε, ασθενών και δείτε τις στατιστικές που έχουν γίνει για τις ε, επιχειρήσεις, τους κλάδους που έχουν ζητήσει κλινικές δοκιμές, θα δείτε ότι δεν είναι μόνο οι φαρμακευτικές εταιρείε, αλλά και ο ακαδημαϊκός κόσμος. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνονται περισσότερο τέτοιες κλινικές δοκιμές, οι οποίες όμως θα τηρούν κάποιες αρχές. Και μιλάω για αρχές γιατί υπήρξαν ε, επικρίσεις που λένε ότι τώρα δεν υπάρχει η υποχρεώση για τέτοιες κλινικές ε, δοκιμές πάντα. Από ό,τι έμαθα, αυτό πορεύει από μια απόφαση υπέρ της στήριξη της αρχής της επικουρικότητας, επειδή στις διάφορες χώρες σήμερα υπάρχουν πολλές καλά οργανωμένες εθνικές επιτροπές που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Ακριβώς λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε την επικουρικότητα και γι' αυτό τελικά δεν ήταν υποχρεωτικό ε, δεν το έκρινε υποχρεωτικό η Επιτροπή Ηθικής να γίνονται τέτοιες ε, κλινικές δοκιμές. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Η πρόταση λέει ότι κάθε χώρα η οποία έχει μηχανισμούς εθνικούς για να, βοηθήσει, να βοηθήσουν μη εμπορική φορείς πρέπει να συμμορφώνεται προς τις αρχές των ε, κλινικών δοκιμών. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη δουλειά, ποιος τελικά θα κάνει τη χρηματοδότηση, Ποιο θα αναλάβει το κόστος. Γιατί εμεί δεν θέλουμε τα κράτη-μέλη να πρέπει να υποχρεωθούν να πληρώνουν. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Μα θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία, όχι να την αυξήσουμε. Συνεπώ, στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τέτοιοι οργανισμοί, όπω αυτοί οι οποίοι αναφέρεται, να μπορούν πιο εύκολα να κάνουν μόνοι του τις κλινικές δοκιμές και ο εντοπισμός εθνικών οργανισμών προβλέπεται στην οδηγία. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω καμία δυσκολία εδώ. Εννοείται ότι πρέπει αυτό να συζητηθεί περισσότερο στη διαδικασία όταν φτάσει στο νομοθετικό επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι τα επίμαχα σημεία που παραμένουν θα διευθετηθούν και εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βοηθήσουμε να πάψουν να υπάρχουν διαφορές που ενδεχομένως υπήρχαν ε, μέχρι τώρα και δυσκολίες που υπήρχαν στην νομοθεσία. Ε, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εγκρίνουμε μέσα στην ε, τρέχουσα εντολή μας. Προτάθηκε τον Ιούλιο του 2012 και συνεχίζονται οι σχετικές εργασίες. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε απόφαση και σε συμφωνία εν ευθέτω χρόνο. Ο πρόεδρος κ. Γκρότε. Επιθυμώ σχετικά με τη διαδικασία να τονίσω και πάλι δεν ε, γνωρίζω μήπως δεν ήσασταν παρούσες ή παρόντες, αλλά η διαδικασία έχει ως εξής. Τίθεται μία ερώτηση και μπορεί να επανέλθει κανείς ως ερωτών εάν θεωρεί ότι η ερώτηση δεν απαντήθηκε πλήρως. Δεν, δεν έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε νέα ερώτηση. Παρακαλώ να σεβαστείτε την ρύθμιση αυτή. Κατρίκα Λεωτάρ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι μπροστά σας. Με βλέπετε. Εφόσον ε, γίνεται επίτροπος, θα έχετε να παίξετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Ευρώπη ολόκληρη δεν θα είναι εύκολο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες ανισότητες ε, όσον αφορά ε, την προσφορά υπηρεσιών υγείας ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Υπάρχει διάκριση σε βάρος των μεταναστών και θα θέλαμε να σας δούμε να δραστηριοποιείτε σε αυτό το τομέα, δηλαδή να φροντίσετε να ενισχύσετε τα δικαιώματα στην υγεία των γυναικών. Και από επιστημονικές έρευνες φαίνεται μέχρι τώρα ότι δεν ε, το ότι δεν ρυθμίζεται η άμβλωση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τεράστιους κινδύνους για την υγεία των γυναικών. Εσείς λοιπόν, ελπίζω ότι θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας, θα φροντίσετε γι' αυτό και θα φροντίσετε για την προστασία ε, της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς στη χώρα σας για παράδειγμα, δεν φροντίσατε να αποφευθούν αυτοί οι κίνδυνοι, στη χώρα σας λέω έτσι, για την υγεία των γυναικών από τις ρυθμίσεις που υιοθετήσατε εδώ. Οπότε πώς θα το κάνετε εδώ τώρα για να μας πείσετε ότι έχετε αξιοπιστία. Πρόεδρος, ένα λεπτό έχουμε, δύο έχει παραπάνω. Να απαντήσει ο Επίτροπος. Όσον αφορά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια συνεκτική πολιτική όπως έχουμε τη συνοχή στα οικονομικά ζητήματα, να τα έχουμε και στην υγεία. Θέλουμε λοιπόν μια πολιτική συνοχής και για την υγεία και τις ανισότητες που υπάρχουν εκεί. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ανισότητες για πολλά σημαντικά θέματα υγείας. Και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μόνο, έτσι. Όσον αφορά την θνησιμότητα των βρεφών, όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, Στη χώρα μου, για παράδειγμα, είμαστε πρώτοι για το προσδόκιμο ζωής. Αλλά αν κοιτάξετε τον χάρτη ανισοτήτων, τότε είναι κάτι που, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ντρεπόμαστε γι' αυτό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι κάτι που δημιουργεί έντονες ανησυχίες. Και βέβαια όταν υπάρχουν ανισότητες πάντα είναι οι πιο ευάλωτοι. Να, στο θέμα το ηλικιακό είναι τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι που υποφέρουν περισσότερο από τέτοιου είδους ανισότητες. Τώρα για το δεύτερο τμήμα της ερώτησή σας να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι θέμα δηλαδή των χωρών μελών να αποφασίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεβαίνει στις αποφάσεις των χωρών μελών, ακόμα και αν θέλει κάποιος δεν μπορεί. Δεσμευόμαστε από τη συνθήκη Υπάρχει το άρθρο 168 της συνθήκης το οποίο διασαφηνίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας είναι στα χέρια των χωρών μελών. Έτσι είναι. Και εγώ συμμορφώνομαι. Είτε μ' αρέσει είτε όχι. Και θα το κάνουμε. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμορφωνόμαστε στο άρθρο αυτό. Πάντως στις χώρες εκείνες όπου οι πρακτικές είναι νόμιμες, ε, συνεχίζουμε. Αν υπάρχει μια άλλη άποψη και σε κάποιε χώρε κάποιε υπηρεσίε είναι παράνομε, ε, θα συνεχίσουν όσο οι χώρε αυτέ επιθυμούν να είναι έτσι. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση? Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο εσείς στη χώρα σας θα δώσετε όθηση σε νέες πρωτοβουλίες στη χώρα σας και τι θα κάνετε όσον αφορά την καταπολέμηση του AIDS, και, του AIDS και την διάδοση των ε, προφυλακτικών, για παράδειγμα, εφόσον μιλάμε για την απαγόρευση της άμβλωσης. Πρόεδρος, έχει δικαίωμα να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ τον υποψήφιο να απαντήσει. Παρακαλώ, ωστόσο, τις και τους συναδέλφους να τηρούν τους κανόνες που οι ίδιοι θεσπίσαμε. Και βεβαίω επίση και τον χρόνο. Οι δεμοί τελευταίοι εγγεγραμμένοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ευγένεια. Οπότε θα απαντήσω κι εγώ ευγενώ. Για την αντισύλληψη βέβαια είναι διαφορετική υπόθεση. Εάν θέλετε, επισκεφτείτε τη Μάλτα και θα δείτε μόνοι σας ότι δεν υπάρχει εκστρατεία κατά της αντισύλληψης. Μάλιστα στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες υπήρχε μια πολιτεία, το Connecticut, που απαγόρευε την αντισύλληψη. Όμω, εδώ δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι πρόκειται για την ελεύθερη επιλογή του κάθε ατόμου. Θα, ήταν, ε, θα αντίκειτο στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο ίδιο το Σύνταγμα τη Μάλτα. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ένα θέμα διάλυση προκαταλήψεων. Η Μάλτα είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω είχε κάποιε παραδόσει ω τώρα, αλλά Δεν ε, ήμουν ποτέ πατριώτη σε βαθμό που να κατεβαίνω στου δρόμου να διαδηλώνω. Θα πρέπει όμω να επειρασπιστώ και την πραγματικότητα της χώρας μου. Για την άμβλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει. Είναι ζητήματα που αποκλειστικώς αποφασίζονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Τώρα, για όσους θέλουν να απελευθερώσουν πλήρως τις πρακτικές αυτές, αυτό είναι το ένα άκρο και υπάρχει και το άλλο που θέλει να τις απαγορεύσει τελείως. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Ευχαριστούμε ο κύριος Σκότα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την δικαιολογία των εξοικονομήσεων χιλιά, ε, ε, εκατομμυρίων ευρώ ετησίως ζητήθηκε από τα ανάλογα λόμπι τις ομάδες πίεσης να αναστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση για την ετικετοθεσία για το βόλιο κρέας με αποκρύπτοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες που απευθύνονται στους καταναλωτές. Εμείς επισημαίνουμε ότι η ευημερία των ζώων και η προστασία του καιρικού περιβάλλοντος είναι προτεραιότητες, αλλά και για την κτηνοτροφία και την επισκεπτική ασφάλεια και την ε, προστασία των καταναλωτών. Έχουμε καταγράψει τι διαμαρτυρίε των Ευρωπαίων ε, κτηνοτρόφων που δεν θέλουν να είναι προαιρετική η ετικετοθεσία στα προϊόντα βόλου κρέατο. Ε, γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πληροφορίε σε ετικέτε, αλλά που να μην είναι απλώ ε, προϊόν φαντασία και να μην ελέγχονται από τι δημόσιε αρχέ. Διότι υπάρχει πολλέ φορέ και βόλιο κρέα το οποίο έρχεται από τρίτε χώρε, εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρέα που πρέπει να ανταγωνιστούν δικοί μα κοινοτρόφοι, που παράγουν προϊόντα ποιότητα. Εσεί λοιπόν, ω υπεύθυνο επίτροπο για τέτοια θέματα, είσαστε υπέρ των κοινοτρόφων και καταναλωτών ή Κύριε Μπόρκ, για, το θέμα της ε, προαιρετικής επικοινωνίας. Ενημερώνομαι ότι η κατάργηση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να επιθέσει την ετικέτα. Απλώς η ετικέτα δεν πρέπει να είναι παραπλανητική στις πληροφορίες που περιέχει. Αυτό το βρίσκω άκρο σημαντικό. Μετά από τη σωρία πληροφοριών που διανέμουμε και συμπεριλαμβάνουμε στις ετικέτες, τελικά ε, βλέπουμε ότι νόημα έχει να μην είναι παραπλανητικές οι πληροφορίες. Οι ετικέτες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό ο οποίος αρχικά έχει οριστεί. Ως Επίτροπος λοιπόν, παρά τη ε, αναστολή του κανόνα που αναφέρατε, θεωρώ ότι η ετικετοθεσία μπορεί να παραμείνει προαιρετική, μπορεί δύναται να γίνεται, αρκεί κανείς να συμμορφούνται με τους κανόνες που ήδη ισχύουν. Δηλαδή να μην παραπλανά τον καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για την εσωτερική αγορά και για τα τρόφιμα και για οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με προϊόντα και εμπορεύματα, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι μια εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών δημιουργεί ένα σοβαρότερο καθήκον για να προστατευτούν οι καταναλωτέ εφόσον δεν υπάρχουν πια εμπορικοί φραγμοί. Υπάρχει, είναι σαν το Σέγγεν. Από τη στιγμή που μπει κανεί, μετά μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο χώρο του Σέγγεν. Σε όλο το χώρο του Σέγγεν. Πολλοί συνηθίζουν να λένε ότι η εσωτερική αγορά βέβαια δημιουργήθηκε για του καταναλωτέ και όχι αντιστρόφω. Έληξε λοιπόν εδώ ο πρώτος γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων και ερχόμαστε στον δεύτερο. Τώρα θα ακολουθήσουν εννέα ερωτήσεις από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα είναι σύντομες ερωτήσεις. Δηλαδή κάθε ερωτών η ε, κάθε ερωτόσα έχει στη διάθεσή της, στη διάθεσή του 50 δεύτερα και ο υποψήφιος έχει στη διάθεσή του για να απαντήσει δύο λεπτά. Παρακαλώ να τηρήσετε αυστηρά το χρόνο διότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Και πρώτη κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, κύριε Μπόρκ. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις ε, υποθέσεις που θα αναλάβετε στο χαρτοφυλάκιό σας, στο πρόγραμμα υγείας πρώτα απ' όλα για το 2014-2020. Η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν θα γίνει αποδεχτή με το Κοινοβούλιο παρά μόνο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι, τα κατάλληλα κονδύλια. Ποια είναι λοιπόν η θέση σα λίγε μέρε πριν ε, τη διάσκεψη κορυφή 22-23 Νοεμβρίου, όταν ξέρουμε ε, ότι δημοσιονομικά τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα. Έπειτα θα φροντίσετε για την καλή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά τη διασυνοριακή υγεία που προβλέπεται για τα τέλη του 2013, ο κύριος Μπόρκ. Ναι, πράγματι. Αυτό είναι ο στόχος μου. Κυρία Κροστέτ, ναι, θα προτιμούσα κι εγώ περισσότερα χρήματα για το πρόγραμμα αυτό υγείας. Έχουμε 64 νομίζω εκατομμύρια για 500 εκατομμύρια καταναλωτές. 2 ευρώ ο καθένας θα το προτιμούσα. Αλλά, εν περιπτώσει, ζούμε τώρα. Και οι προτάσεις μας και τα προγράμματά μας πρέπει να προετοιμαστούν και οι πρωτοβουλίες μας υπό το φως της πραγματικότητας που έχουμε. Ξέρω ότι υπάρχει τριμερής διάλογος αυτή την εποχή και να ξέρετε ότι εγώ θα σταθώ πολύ κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο γιατί αυτό είναι το πιο ε, βολικό, αλλά γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί αυτό θέλει ο κόσμος. Εσείς είσαστε ο δημοκρατικός βραχίωνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι κοινοβουλευτικό επειδή ε, τυχαίνει να ε, ανήκω σε ένα σύστημα που για να γίνει κανείς υπουργό πρέπει να είναι κοινοβουλευτικός, βουλευτής. Αλλά εσείς εκπροσωπείτε τους λαούς των χωρών σας εσείς ξέρετε ποιες είναι οι προτερότητές τους και πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου για το πρόγραμμα υγείας, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε έτσι ώστε τα συστήματα υγείας να είναι πιο σταθερά, που υπάρχουν ε, ανισότητες, να τις αντιμετωπίσουμε. Επίσης να δούμε και το θέμα της καταπολέμησης των χρόνιων ασθενών. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον παράγοντα κινδύνου ή την διατροφή, την κατανάλωση αλκοόλ, ή καπνού, η έλλειψη ε, σωματικών ε, δραστηριοτήτων, άσκησης. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ως παράγοντες κινδύνου, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ο χρόνος να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί, αλλά και με άλλους για να προχωρήσουμε. Σίγουρα και αυτό θα το προσέξω κυρία Γκροστέτ. Κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ, παιδε. Κυρία Μπόρκ, οι προσωπικές σας πεπιθήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και την άβλωση είναι γνωστές. Στην ακρόαση αυτή αρνηθήκατε στο όνομα της αρχής της επικουρικότητας να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις που σας έφερναν σε δύσκολη θέση. Κύριε Μπόρκ, τι εγγυήσει αμεροληψίας και ανεξαρτησίας μπορείτε να μας προσφέρετε. Όχι μόνο ως Επίτροπος Δημόσιας Υγείας, αλλά και ως μέλος του Κολεγίου Επιτρόπων όταν θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Όχι μόνο των γυναικών της Ευρώπης, αλλά και των γυναικών των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό ζητούμε να μάθουμε και εδώ θέλουμε συγκεκριμένη και σαφέστατη απάντηση. Ευχαριστώ. Κύριε Μπόρκ. Αλήθεια είναι ότι είμαι δικηγόρος αλλά δεν ψάχνω και καταφύγιο και να αποφύγω τι απαντήσει. Οι συνθήκε πρέπει να εφαρμοστούν. Το αν συμφωνώ ή όχι είναι τελείω διαφορετικό. Πρέπει να εφαρμοστούν οι συνθήκε και είναι σαφεί οι συνθήκε για τα θέματα που αναφέρατε. Απήντησα ειλικρινέστατα και πολύ ανοιχτά. Δεν θα εγκαταλείψω τι προσωπικέ μου απόψει. Θα ήταν υποκριτικό κάτι τέτοιο. Και θα το καταλαβαίνετε και αμέσω εάν το είχα αποπειραθεί. Αυτό που υπόσχομαι είναι ότι θα συμμορφωθώ με την περιγραφή των καθηκόντων μου εφόσον περάσω τη διαδικασία. Πρέπει να συμμορφωθεί κανείς με τους κανόνες της ομαδικότητας, διότι ε, ιδάλλως θα είχαμε 27 επιτρόπους, όχι μία ενιαία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανόνας, ε, η αρχή της επικουρικότητας, δεν επιτρέπει να ακολουθήσουμε τις πρακτικές της πλειοψηφία των κρατών μελών. Το αντίστροφο συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε προγράμματα ή στην νομοθεσία χωρών που είτε είναι η πλειοψηφία είτε όχι ασκούν συγκεκριμένες πρακτικές. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να παρέμβω. Πρώτον γιατί δεν θέλω, δεύτερον γιατί δεν έχω το δικαίωμα και τρίτον γιατί θα παραβίαζα όσα ορίζουν οι συνθήκε αν το έκανα αυτό. Και δεν έχω και καμία εντολή να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ψάχνω να αποφύγω απαντήσεις, απλώς σας αναφέρω τι λένε οι ίδιες οι συνθήκες. Ορκίζομαι να είμαι ε, Ευρωπαίος Επίτροπος. Στην ε, προσωπική μου ζωή ε, και με τις προσωπικές μου πεπιθήσεις, όσο και αν άλλαζα ιδιότητες επί 30 χρόνια, πολέμησα για να προσχωρήσει η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για τα κονδύλια και τις επιδοτήσεις, αλλά για να προσαρτήσει, να προσαρτήσει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο ενδιαφέρον μια περιφερειακή χώρα να βρει αγκυροβόλιο στο κέντρο, στο λιμάνι του κέντρου της Ευρώπης, στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές που συμμεριζόμαστε, γιατί και εμείς είμαστε μέρος αυτής της Ευρώπης. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμαινε ακριβώς αυτό. Να ε, περάσει για πάντα στο λιμάνι των ευρωπαϊκών αξιών η Μάλτα ο Πρόεδρος. Θα απευθύνω έκκληση στους προσκεκλημένους που κάθονται στο πίσω μέρος του αίθουσας. Δεν βρισκόμαστε εδώ ούτε σε συναυλία pop ούτε στο γήπεδο. Είτε επιδοκιμαστικά είτε αποδοκιμαστικά σχόλια, παρακαλώ, δεν έχουν καμία δουλειά να προέρχονται από τους προσκεκλημένους. Παρακαλώ ασκήστε κάποια αυτοπιθαρχία ώστε να μπορέσει η διαδικασία να εξελιχθεί μέσα σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο. Ο κύριος Πέτερλε, Αλόης Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε υποψήφιε. Θα ήθελα να σας υποβάλω μια ερώτηση η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων σας. Γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος αναπτύσσεται στους ασθενείς πολύ ταχύτερα από ό,τι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε πώς μπορείτε να βελτιώσετε τον αγώνα κατά του καρκίνου στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τι προληπτικές δράσεις σκοπεύετε να αναπτύξετε. Άκουσα με ενδιαφέρον τις αρχικές σας δηλώσεις, καθώς επίσης και για θέματα ασφάλειας τροφίμων, όπου βάλατε βεβαίως την αρχή της ασφάλειας πριν από την αρχή της ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ κύριε Μπόρκα, έχετε το λόγο. Υπάρχει έστω και μία οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην έχει στους κόλπους της κάποιον που επλήγει από τον καρκίνο, πιστεύω πως όχι. Εγώ και στη δική μου οικογένεια έχω ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν από την ασθένεια αυτή. Και βεβαίως η πρωταρχική τάση θα πρέπει να είναι, όχι βεβαίως να αντιμετωπιστεί η ασθένεια αφήσει διαγνωστή, και αυτό είναι σημαντικό βέβαια, αλλά να γίνει προσπάθεια πρόληψης. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, υπάρχει μεγάλος αριθμός καρκίνων που μπορεί να προληφθεί. Αν εξετάσουμε τους προϋπολογισμούς των εθνικών συστημάτων υγείας, θα δούμε ότι το 3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης πηγαίνει στην πρόληψη και 97% στην θεραπεία. Θα είναι δύσκολο να αλλάξει αυτή η αναλογία, αλλά πάντως πρέπει να βελτιωθούν τα νούμερα αυτά και για την ασθένεια που αναφέρατε, ειδικότερα το πιο σημαντικό πρόγραμμα που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει η ΣΑΝΚΟ και οι υπηρεσίε μου θα είναι η ενθάρρυνση πέραν από τις εκστρατείες ενημέρωσης η ενθάρρυνση του screening της πρώτερης δηλαδή εξέτασης όπου γνωρίζω και από την πατρίδα μου ότι πολλές ζωές έχουν σωθεί από την πρόορη διάγνωση των καρκίνων του μαστού. Καθώς και τα γενικά που ανέφερα προηγουμένως, ο αγώνας δηλαδή κατά των χρόνιων ασθενειών, χρόνιων νόσων, όπως διαβήτης, καρδιαγκιακά και καρκίνος, που είναι και οι πιο σημαντικοί, ε, οι πιο σημαντικές μάλλον αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως ταυτόχρονα με την βελτίωση των διατροφικών συνηθιών, μείωση του καπνίσματος κλπ. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Μπορούν ωστόσο να θεσπιστούν τέτοιοι στόχοι ώστε να μειωθούν και να μειωθεί και η συχνότητα εμφάνιση του καρκίνου. Ζιλ Πανιό. Κύριε υποψήφια, είπατε ότι επιθυμείτε να είστε επίτροπος που θα διακριθεί για την ειλικρινιά του. Θα σας ρωτήσω για ένα θέμα που νομίζω απαιτεί κάποια διαφάνεια και μάλιστα περισσότερη διαφάνεια από τον προκάτοχό σας. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων δηλαδή που εγώ θεωρώ ότι απειλείται σήμερα από τις συγκρούσεις συμφερόντων. Δημοσιεύεται έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την σύγκρουση συμφερόντων σε τέσσερις οργανισμούς της Ένωσης, δύο μάλιστα που θα εμπίπτουν και στο χαρτοφυλόγιο σας και που λέει ότι κανένας από τις ελεγχθέντες οργανισμούς δεν έχει χειριστεί με σωστό τρόπο τις συγκρούσεις συμφερόντων. Ερώτηση λοιπόν, πώς θα προβείτε σε βαθιά αναμόρφωση των οργανισμών σε εφαρμογή των συμπερασμάτων της εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου με δύο συγκεκριμένα πράγματα για το μπισφενόλ α και για, την, για το ασπαρτάμ και με τον τρόπο αυτό θα απαντήσετε και στην ανησυχία του συνάδελφου Πέτερλε για τον καρκίνο. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας που νομίζω ότι πράγματι έχει άκρα προτεραιότητα. Και άκρα προτεραιότητα λέγω διότι την υγεία εργάζονται δύο σημαντικοί ανεξάρτητοι οργανισμοί, η ΕΦΣΑ στην Πάρμα και η Βέρμα στο Λονδίνο. Γνωρίζω καλά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για έναν ολόκληρο αριθμό ανεξαρτήτων οργανισμών. Η έκθεση αυτή εντοπίζει σφάλματα σε όλους τους οργανισμούς αυτούς. Ίσως αυτό να παρηγορεί ορισμένου, την ΣΑΝΚΟ δηλαδή. Η ΕΜΑ και η ΣΑΝΚΟ ήταν από τους οργανισμούς εκείνους που είχαν τα λιγότερα σφάλματα. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτη παρηγοριά. Εγώ θα συμμορφωθώ με τις συστάσεις της εκθέσεως του ελεκτικού συνεδρίου. Και ιδιαίτερα διότι η ΕΦΣΑ και η ΕΜΑ όχι μόνο πρέπει να είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί, αλλά και πρέπει να γίνονται αντιληπτοί ως ανεξάρτητοι. Καμιά φορά η αντίληψη που έχει κανείς ε, είναι το ίδιο σημαντική όπως και η πραγματικότητα στα, ε, στα πολιτικά. Ωστόσο, α διατηρήσουμε τους οργανισμούς αυτούς, σας μην του αμαυρώσουμε, διότι δεν είναι προ το συμφέρον μας να τους αμαυρώσουμε. Είπα προσφάτω σε κάποιον ότι από τη στιγμή που η ΕΦΣΑ θα γίνει δημοφιλής, εγώ θα αρχίσω να ανησυχώ. Διότι είτε θα επικρίνεται διότι είναι πάρα πολύ αυστηρή, όπως με τους ισχυρισμούς ε, υγείας, τα health claims, είτε διότι είναι πολύ επίκη. Και η σωστή πορεία βέβαια είναι κάπου ανάμεσα. Έτσι λοιπόν, ναι, θα επιβάλλω μέτρα για την εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις συμφεράντων και ιδίως σε ό,τι αφορά πρακτικές μετά την απασχόληση, αλλά και διότι θεωρώ ότι και με άλλους βέβαια συναρμόδιους επιτρόπους θα πρέπει να θεσπίσουμε κοινού κανόνες για την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων για όλους τους οργανισμούς και όχι μόνο για έναν. Ο κάθε ένας θα έχει βέβαια τις ιδιαιτερότητές του. Ωστόσο, χρειαζόμαστε κάποιου κοινού κανόνε. Βέβαια, αυτό δεν εξαρτάται μοναχά από μένα. Αυτή είναι βεβαίω η προσωπική μου άποψη, την οποία σα μεταφέρω. Η κυρία Οκονή, 50 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφια, καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εργάζομαι στην Επιτροπή αυτή ιδιαιτέρως για τα θέματα τα, ε, των τροφίμων. ω προ την ετικετοθεσία του βοήου κρέατος. Ήθελα να μας πείτε ποια η δική σας θέση για την κλωνοποίηση ζώων με σκοπό την ε, παραγωγή τροφίμων. Από την εισήγησή σας ακούσαμε ότι θα υποβάλλετε μια πρόταση του χρόνου. Δώστε μου κάποιες λεπτομέρειες για τη δική σας την τοποθέτηση σε σχέση με το θέμα αυτό. Θα ξέρετε ότι το Ευρωκοινοβούλιο παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το όλο ζήτημα. Έπειτα, από την ε, θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχει αρμοδιότητα και για, την, ε, για τον αθλητισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθοριστική σημασία για σκοπού δημόσια υγεία. Θα πρέπει να μπει στο κέντρο τη ε, πολιτική αυτή. Τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά, κύριε Μπόρκ. Για την κλωνοποίηση ζώων, προείπα ότι θα υποβάλουμε και θα προωθήσουμε πρόταση ώστε ως τον Ιούνιο του 2013 να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν όλα πάνε καλά, μια οδηγία και για την κλωνοποίηση και για τα νέα τρόφιμα. Γνωρίζουμε το ιστορικό της τελευταίας πρότασης. Ας διδαχτούμε από το παρελθόν. Δεν θέλω να την αποκαλέσω σφάλμα, ας την αποκαλέσουμε εμπειρία. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που να απαγορεύει την κλωνοποίηση με σκοπό την παραγωγή τροφίμων. Δεν το βρίσκω σωστό αυτό. Νομίζω ότι η αναπαραγωγή ζώων για, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, αυτή ακριβώ τη στιγμή, σήμερα, δεν έχουμε τέτοιο νόμο. Γιατί, α αναρωτηθούμε γιατί. Γνωρίζουμε τι συνέβη όταν έγινε η πιο πρόσφατη απόπειρα. Πρέπει να κάνουμε ένα νέο βήμα πλέον, ώστε η κλωνοποίηση των ζώων να απαγορευτεί επιτέλου. Το πρόβλημα βέβαια δεν θα προκύψει σε αυτόν τον χώρο. Ούτε νομίζω στο Κοινοβούλιο και ούτε και στο Συμβούλιο. Σε άλλου χώρου θα προκύψει. Με την ετικετοθεσία των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα, ε, για την γενιά από την οποία θα πρέπει να επιβάλλεται και μετά. Βεβαίω με αυτό θα πρέπει να, γι' αυτό θα πρέπει να συνοηθώ και με άλλου επιτρόπου, διότι επικαλύπτονται και άλλοι τομεί, αλλά είναι θέμα δημόσια υγεία και σκοπεύω να προωθήσω την πρόταση αυτή υγεία, ώστε να εγκριθεί ω τον Ιούνιο του 2013. Για τα νέα τρόφιμα δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Για τον αθλητισμό, μείωσα την ε, σημασία της άσκησης, της φυσικής, της φυσικής Τη σωματική άσκηση για σκοπούς δημόσια υγείας. Στο βαθμό λοιπόν που μπορούμε, ε, εγώ και οι υπηρεσίε μου θα προωθήσουμε τον αθλητισμό, κυρίω μεταξύ των νέων, αλλά κρίνοντας και την προσωπική μου εμπειρία, ποτέ δεν είναι αργά. Ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει μια αθλητική δραστηριότητα. Το προτείνω στον καθένα στην αίθουσα αυτή. Ε, Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε τα θέματα υγείας και την ε, αξίωση αποζημιώσεων για θέματα υγείας. Δεν ε, υπάρχει συμφωνία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δεν το πετύχαμε το 2006. Αν ε, όμως αυτό γίνει για προϊόντα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, Έπειτα, πολλές φορές, και εδώ πέρα μιλάω περισσότερο για τους ισχυρισμούς ότι ορισμένα προϊόντα έχουν κάποιες συγκεκριμένες συνέπειες στον οργανισμό. Πώς θα προστατεύσουμε και κυρίως τους γονείς για ισχυρισμούς που κάνουν οι γαλακτοκομικές εταιρείες ε, για τα γάλατά τους. Πώς θα προχωρήσετε με αυτό το θέμα για το γάλα για τα νεογνά. Όπως έχω ήδη πει, αυτό είναι ένας τομέα όπου έχει επικριθεί πολύ εύσα. Και γιατί? Γιατί όταν γίνονται ισχυρισμοί για επιπτώσεις στην υγεία από εταιρείε τροφίμων, ε, διαπιστώσαμε ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το οποίο ισχυρίζονταν. Εμείς δεν απαγορεύουμε κάποια τρόφιμα με τη ρύθμισή μας, απλώς προσέχουμε να μην υπάρχουν ψευδείς ισχυρισμοί. Βλέπετε μερικές φορές έχει επικριθεί η Εύσα για αυτά που κάνει, σαν έχει απαγορεύσει κάποια τρόφιμα. Όχι, δεν απαγορεύει τα τρόφιμα αυτά, λέει απλώς ότι αυτός ο συγκεκριμένος ισχυρισμός ότι βελτιώνει τη χώνεψη ή ότι σας βοηθάει να δυνατήσετε, ε, δεν ισχύει. Και ο καταναλωτής πρέπει να το ξέρει αυτό, δεν πρέπει να ξαπατάτε. Όσον αφορά τώρα το διατροφικό προφίλ, εγώ κάνω αυτό που λέει ο νόμος. Η νομοθεσία έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια πρέπει και να τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά δεν είναι ότι τώρα φτιάχνουμε καινούρια νομοθεσία. Όχι, πρόκειται για την εφαρμογή μιας νομοθετικής ρύθμισης η οποία περιμένει να εφαρμοστεί ακριβώς. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη διαδικασία και τα παραδοσιακά τρόφιμα, να τα προστατεύσουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Και ο λόγος είναι ότι Πάντα μπορεί κάποιο να προβάλλει ψευδείς ισχυρισμού λέγοντας ότι το συγκεκριμένο τρόφιμο βοηθάει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη πτυχή της υγείας, αλλά ελοχεύει κινδύνους για κάποιο άλλο, κάποια άλλη πτυχή της υγείας. Ε, αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, με αυτήν ακριβώς τη ρύθμιση για το προφίλ των τροφίμων. Ευχαριστώ. Είχαμε και μια δεκαετία επέτειο πολύ σημαντική πέρσι για την ε, Επιτροπή μας. Τώρα η κυρία Αντωνέσκου, 50 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είστε παρόν κύριε υποψήφια Επιτροπέ. Έχουμε μια οικονομική κατάσταση ιδιαίτερα δυσχερή. Σε πολλές χώρες υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες και χρειάζεται να γίνει συνεργασία και για την ιατρική ε, παρακολούθηση και παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών. Οι ε, πολίτες πιστεύουν ότι υπάρχει άνηση μεταχείριση και αυτό και για χρόνιες παθήσεις. Άκουσα τα όσα είπατε για τις ελλείψεις ισότητας. Χρειαζόμαστε μια συνοχή, όπως είπατε και εσείς, και στον τομέα της υγείας, όπως και για τα οικονομικά. Έχω εδώ μια ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω, εάν προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις ανισότητες αυτές, και να προσφέρετε ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και αν αυτό θα το καταστήσετε προτεραιότητά σας. Κύριε Μπόρκ, έχετε το λόγο. Ναι, βεβαίως θα αποτελέσει μια από τις προτεραιότητές μου, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με διάφορες ιδέες, όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, όπως ενότητα μέσα στην ποικιλία. Αλλά πρέπει η πολυφωνία. Πρέπει όμως να μην λησμονείται και η αρχή τη αλληλεγγύη. όχι βεβαίως να εγγράφεται στα εγχειρίδια ή στις διακηρύξεις, αυτό είναι εύκολο, αλλά και να εφαρμόζεται σε διάφορου τομεί. Αλληλεγγύη επίση σημαίνει και στον τομέα της υγεία. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το τι θα πρέπει, για το πού θα πρέπει να κατευθύνουμε τις προσπαθίες μας. Όσον αφορά συγκεκριμένες δράσεις, έχω μία υπόψη μου, ξεκάθαρα, την υποστήριξη δηλαδή, τις, τα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεως για τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν λιγότερο το 90% του GNI και να κάνουμε διάκριση υπέρ αυτών. Η διάκριση δεν μπορεί να απαγορεύεται πάντοτε, γιατί υπάρχουν φορά και θετικές διακρίσεις. Για το 90% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτά λοιπόν, αυτέ οι θετικέ διακρίσει πρέπει να ισχύουν και στον τομέα τη υγεία. Όσοι χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη πρέπει να την λαμβάνουν. Διάκριση που δεν αποτελεί πράγματι διάκριση, διότι αυτή τη στιγμή είναι θετική, δεν μπορεί καν να οριστεί ω διάκριση. Πρόκειται αλληλεγγύη. Μεταμορφώνεται από διάκριση σε αλληλεγγύη. Αυτό είναι ένα από τα προγράμματα που θα ήθελα να προωθήσω την συγχρηματοδότηση δηλαδή. Ίσως να μην συμφωνούν όλοι βέβαια μαζί μου, αλλά πιστεύω ότι όσοι χρειάζονται την υποστήριξη αυτή για θέματα υγείας θα είναι υπέρ. Και ας μην λησμονούμε επίσης ότι οι φτωχοί έχουν δικαίωμα και αυτοί στην υγεία. Η φτώχεια σημαίνει και ευάλωτο. Σας ευχαριστώ, Λέω Πρόεδρος. Και βάλω τη βεβαίω και λόγω, ε, μπορεί και λόγω ηλικία. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, λέει ο κύριο Σνέλχαρτ, για την πολιτική 2007 έως 2013 μιλούμε και για την υγεία ανθρώπων αλλά και ζώων. Και έχουμε τη στρατηγική για την υγεία των ζώων που έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποιοι ότι θα προωθηθούν κανόνες για την κτηνιατρική συνεργασία κλπ. Ωστόσο οι προτάσεις αυτές δεν έχουν κατατεθεί. Το 2013 λίγη η φάση αυτής της στρατηγικής. Θεωρείτε ότι το θέμα αυτό πρέπει να γίνει επίκαιρο. Γιατί έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και γιατί η Κομισιόν θα υποβάλει και θα υποβάλει η Κομισιόν ένα πακέτο με όλες αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπόρκ. Η πρόθεση της δέσμης μέτρων είναι να υποβληθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Θα συνενώσει τα όσα ήδη έχουν υποβληθεί σε ένα ενίο πακέτο. Μιλώντας χωρίς προετοιμασία θα έλεγα ότι για θέματα τα οποία απασχολούν όλους, ιδίως για την αντίσταση στα αντιβιωτικά στην, στον τομέα της υγείας των ζώων, που βεβαίως επηρεάζει και την υγεία των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πραγματικά αν όντως επιβάλλουμε την ισχύουσα νομοθεσία, διότι δίνοντας αντιβιωτικά σε ανθρώπους ή σε ζώα, όταν κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, σημαίνει ότι μειώνουμε την ανθεκτικότητα των οργανισμών τους, κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο για ε, τους ίδιους, για την υγεία των ζώων δηλαδή, αλλά και την ε, αύξηση της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά έχουν ένα κύκλο ζωής και εν τέλει επηρεάζεται αυτός ο κύκλος ζωής, αλλά με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται και η φαρμακευτική βιομηχανία. Διότι επενδύει βεβαίω η φαρμακευτική βιομηχανία βεβαίω για λόγου κέρδου σε ένα αντιβιωτικό με πρόβλεψη κάποια χρονική περίοδου. Τώρα όμω αυτή η χρονική περίοδο μειώνεται τόσο πολύ που καταστρέφει ακόμη και την κερδοφορία τη βιομηχανία. Που είναι απαραίτητο να υπάρχει ωστόσο για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε έρευνε για την παραγωγή νέων αντιβιωτικών. Άρα η δέσμη αυτή μέτρων βρίσκεται στο λεγόμενο pipeline, στον αγωγό, έρχεται λοιπόν και ελπίζω ότι θα ενισχύσει και τις ε, αρμοδιότητες ή τις εξουσίες επιβολής και όχι, που διαθέτουμε όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα των αντιβιωτικών αλλά και για άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, των φυτών και των σπόρων. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους σπόρους διότι και οι σπόροι μπορούν να προκαλέσουν ε, ολόκληρη αλυσίδα ε, μολύνσεων από γενιά σε γενιά σπόρων. Ο κ. Γκρίφιν δεν είναι παρόν. Τότε λοιπόν έληξε εδώ ο δεύτερος γύρος των ερωτήσεων. Και θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις της Επιτροπής Ενιαίας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών και εδώ θα αναλάβει τα, τη διεύθυνση της συζητήσεως ο κύριος Χάρμπορ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ εξ ονόματος των μελών μας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος που μας προσφέρει την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε με τον υποψήφιο επίτροπο κρίσιμα θέματα του χαρτοφυλακίου του. Υπενθυμίζω στις και στους συναδέλφους μου ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουν, να θέσουν οι συναδέλφοι μου δηλαδή 7 μακρές ερωτήσεις, ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η ε, απάντηση και μετά ενδεχομένως συμπληρωματική ερώτηση. Μετά θα έχουμε τρεις βραχίες ερωτήσεις και εισαγωγικά βεβαίως γνωρίζω ότι θα παρακολουθούν πολύ, πολύ προσεκτικά το χρονόμετρο οι συναδελφοί μου της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση τον υποψήφιο επίτροπο στην εισαγωγική του ομιλία να λέει ότι θα ηγηθεί της προσπάθειας προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ενέργειας αγοράς. Αυτά είναι τα θέματα που γνωρίζω ότι θα θέσουν ως ερωτήσεις και οι συναδελφοί μου. Θα αρχίσω λοιπόν δίνοντας το λόγο στον κύριο Σβάπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ακριβώ εκεί ήθελα να έλθω και εγώ κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Στην εισαγωγική σας ομιλία είπατε ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, να γίνουν πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, πώς θα επιτύχουμε η εγκεκριμένη νομοθεσία να υλοποιηθεί, να επιβληθεί στις χώρες μέλη και τέλος για να εφαρμοστεί με ισότιμο τρόπο σε όλες τις καταναλώτες και τους καταναλωτές. Δεύτερο, υπάρχει πρόσφατη μελέτη που δείχνει ότι πολλές καταναλώτρες και καταναλωτές συχνά δεν είναι εις θέση να κατανοήσουν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους παραγωγούς. Θεωρείται ότι είναι δυνατόν να ενημερωθούν με κατάλληλο και σκόπιμο τρόπο οι καταναλωτές. Ευχαριστώ. Κύριε Μπόρκ. Είναι πολλά τα εργαλεία που διαθέτουμε. Το θέμα είναι αν τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά, σωστά και αποδοτικά ή όχι. Εάν δεν είμαστε αυστηροί στην επιβολή, αυτό θα είναι άδικο και για τους καταναλωτές, αλλά και όσους συμμορφώνονται με τους κανόνες. Εάν δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ σεβασμού των κανόνων και μη σεβασμού, του, σεβασμού τους, ε, όλοι δεν θα τους σέβονται. Πρόκειται για κανόνε που μέσα από την διαδικασία τη συναπόφαση του έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια διαδικασία που την έχω μελετήσει στο παρελθόν, τώρα έχω και άμεση εμπειρία της. Είναι λοιπόν κάτι που θα ισχύσει αυτό για όλη την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν σοβαρές ε, διαφορές. Σκοπεύω να παραστώ στη σύνοδο αυτή, στη σύνοδο κορυφής των Υπουργών που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών με θέμα την επιβολή. Βεβαίω, δεν μπορούν να επιβληθούν όλοι οι νόμοι ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο και χωρί εξαιρέσει. Είναι ανέφικτο. Αλλά πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας και διαθέτουμε εργαλεία στη διάθεσή μα. Έχουμε το κέντρο προστασία των καταναλωτών που έχουν ε, συντονίσει τις προσπάθειες των ενώσεων καταναλωτών, αλλά και για τα ένδικα μέσα. Μέσα από την νομική μου εμπειρία, έχω εργαστεί 15 χρόνια ως δικηγόρος, ακριβώς στα δικαστήρια, στην ίδια την αρένα της ε, νομικής επιστήμης, ε, με την επίλυση διαφορών και την εκδίκαση υποθέσεων. Το να λέει κανείς στον καταναλωτή ότι μπορεί να προσφύγει, είναι πολύ ωραίο επί χάρτου, αλλά στην πράξη μοιάζει με στιγματισμό για κάποιους. Το να μπουν σε ένα δικαστήριο ακόμα. Πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε νέες μεθόδου. Υπάρχει σχετική νομοθεσία σε επεξεργασία, όπου ένα καταναλωτή θα μπορεί να προσφύγει για κάτι με λιγότερο δαπανηρή διαδικασία, με εναλλακτική διαδικασία και με ταχύτερε εκδικάσει υποθέσεων. Διότι εάν με ρωτήσετε ποιε είναι οι προτεραιότητέ μου για τον καταναλωτή, είναι η ασφάλεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση αλλά και η επιβολή. Αυτέ είναι οι τέσσερι προτεραιότητε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει και την εκπαίδευση των καταναλωτών στο ίντερνετ, ε, διαδικτυακά για τα ταξίδια, για την αγορά εμπορευμάτων διασυνοριακά. Θα πρέπει λοιπόν ε, στο μέλλον να βελτιωθούν όλε αυτέ οι υπηρεσίε που θα αναλωθεί. Συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Σφάμπ. Συμπληρωματική. Αυτό σημαίνει όμως ότι σε ορισμένες διασυνοριακές περιστάσεις θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια εναρμόνιση των δικαίων των καταναλωτών, διότι η προστασία της οποίας χαίρουν οι καταναλωτές σε διαφορετικές χώρες είναι διαφορετική. Ποια βήματα προτίθεστε να λάβετε σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Στην πρώτη μου ε, παρέμβαση δεν αναφέρω πίνακα βαθμολογία, λόγου χάρη. Για του ε, καταναλωτέ είναι κάτι βέβαια που δεν είναι πολύ γνωστό και πολλέ φορέ επικρίνεται γιατί θεωρείται δαπανηρό. Όμω είναι μία μέθοδο όχι μόνο για να βαθμολογήσει κανείς τις δικές του επιδόσεις, αλλά να μπορεί και κάποιος άλλος να μάθει ποιες είναι οι επιδόσεις σου. Να το ονομάσουμε πονηδισμό. Ε, εγώ νομίζω ότι πιο σωστό θα ήταν να λέμε ότι κατονομάζουμε και βάζουμε στη σωστή ιεραρχία. Παρά επονηδίζουμε. Βεβαίω, αν βρίσκεται κανεί στο κάτω-κάτω μέρο τη βαθμολογία, είναι αυτό αρκετά στενάχωρο. Όμω, οι πολιτικές κυρώσεις είναι εξίσου σημαντικές όπως και οι νομικές. Άρα υπάρχουν τρόποι και μέσα να ενδυναμωθεί η επιβολή. Πρέπει να τα επιχειρήσουμε όλα αυτά. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα σημαντικά των καιρών. Εάν δεν το κάνουμε όλο αυτό, όλες μας οι προσπάθειες δεν καταρρεύσουν. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος για την εσωτερική αγορά. Μια αγορά με 500 ε, ε, εκατομμύρια καταναλωτές. Εάν ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές, μπορεί να κυκλοφορήσει μεταξύ 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και τώρα η κυρία Γκέπχα, την οποία καλωσορίζω θερμά στην ακρόαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, στον πρώτο γύρο απαντήσατε συχνά με αναφορά σε σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και με την επίκληση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων καταφέρατε να μην απαντήσετε. Τώρα έχω ερωτήσει. Η κυρία Ρέντινγκ προτίθεται να καταθέσει πρόταση νομοθεσίας για ορισμένα θέματα. Θα την ενισχύσετε ή όχι στο συλλογικό όργανο των Επιτρόπων. Δεύτερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό για κάθε πολίτη ανεξαρτήτως φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας το υποσχέθηκαν αυτό, αλλά δεν βλέπω για την ώρα τίποτα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν γίνεται επίτροπος, θα υποστηρίξετε τον κύριο Μπαρνιέ για να προχωρήσει σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, ναι ή όχι. The, the, the η ερώτηση. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να απαντήσω, αλλά δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητα της συγκεκριμένης επιτροπής, παρόλα αυτά ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε την απάντησή σας. Κοιτάξτε, δεν θα αποφύγω, η απάντηση είναι ναι και ναι. Δεν θα χρονοτεπίσω. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Βεβαίω δεν θα σταματήσω εδώ. Να αναπτύξω γιατί απαντάω καταφατικά. Ναι και ναι για τις ποσοστώσεις είναι κάτι που ορίζεται από, τις, από τη χάρτα. Απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου και ε, αλλά για κάποιες ειδικές περιπτώσεις υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν έχω λοιπόν πρόβλημα με τις ποσοστώσεις, αλλά θα πρέπει κανείς να δει τις λεπτομέρειες της ίδιας της πρότασης, γιατί πολλοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τις ε, θέσεις των ερέσιμων ε, λειτουργών, αλλά όχι για τα αριθμιστικά σώματα, λόγω χάρη, για τις τραπεζικούς λογαριασμούς. Νομίζω ότι το είχα ήδη καλύψει στην αρχική μου συζήτηση, μια υπόσχεση. Η πρόταση θα υποβληθεί, όμως θα πρέπει να το δω περαιτέρω με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον καθέναν. Διότι πραγματικά θα αλλάξει πολλά για τον κάθε καταναλωτή. Δεν είναι κάτι ασαφές και θεωρητικό. Είναι κάτι που θα επηρεάσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων γυναικών και ανδρών ε, γύρω μας. Περισσότερη διαφάνεια, δυνατότητα καλύτερης γνώσης για τους δασμούς που επιβάλλονται Από ό,τι γνωρίζω από τι υπηρεσίε μα, ήδη το Φεβρουάριο του 2013 θα είναι έτοιμη διαδικασία έγκριση. Συμπληρώσει. Για αυτό το δεύτερο θέμα, μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, όχι πλέον για τη διαφάνεια ή την αλλαγή λογαριασμών, αλλά για τη φροντίδα ώστε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Στι απαντήσει σα μέχρι τώρα έχετε μιλήσει μονάχα για πρωτοβουλίε. Αυτό το βρίσκω ασαφέ, αόριστο. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα. Ε, ενάξιμο δικαίωμα, δηλαδή ένα δικαίωμα για το οποίο να μπορούν να προσφύγουν κιόλα οι καταναλωτέ για την πρόσβαση σε λογαριασμού. Απάντηση. Συμφωνώ. Πρόκειται για προσβασιμότητα σε λογαριασμό, διότι εν τέλει ο λογαριασμό έχει γίνει το ίδιο απαραίτητο για τον καθένα όπω και η ταυτότητα, διαφάνεια για τα τέλη που πληρώνει κανεί και το θέμα τη δυνατότητα αλλαγή λογαριασμών. Ο τίτλο τι οδηγίε θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να γίνει ένα αυτοδύναμο δικαίωμα. Ευχαριστώ. Μάντερς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπόρχ, ασχολούμαστε με την προστασία των καταναλώτων. Είμαι καταναλώτης και εγώ. Και πιστεύω ότι πρέπει να με προστατεύσετε και εμένα. Ο κύριος Δελή έπρεπε να φύγει για μια υπόθεση που προέκυψε, ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα έχετε μια πάρα πολύ σημαντική θέση και ότι η Όλαφ πάντα θα είναι εδώ για να ελέγχει. Ο κύριος ε, Νταλή ήταν υπέρ της ε, πρόληψης στην ε, υγεία. Ελπίζω να είσαστε κι εσείς υπέρ της πρόληψης στην υγεία. Και για να υπάρχει τέτοια πρόληψη πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τις σωστές επιλογές στα τρόφιμα που τρώμε. Και αυτό ισχύει για τους νέους. Οπότε εσείς πώς θα φροντίσετε να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες οι καταναλωτές ασθενείς, αλλά και στις κατάλληλες θεραπείες και στα κατάλληλα φάρμακα. Ούτε αυτά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, αλλά εν πάση περιπτώσει για την πρώτη ερώτηση το θέμα της Όλαφ δεν έχει να κάνει εδώ με την ε, Επιτροπή μας, αλλά ο κύριος Μπόρκο θα απαντήσει όσο πιστεύει ότι θέλει να απαντήσει σε αυτά. Μα το θέμα δεν είναι πόσο ευφύς είναι κανείς. Γι' αυτό το θέμα ήρθα σε επαφή με το γραφείο του κύριου Νταλή και ελπίζω ότι θα έχει στη διάθεσή του ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υπήρξε μια παρέτηση και μια αντικατάσταση έρχεται. Η κυβέρνησή μου με πρότεινε να αντικαταστήσω τον κύριο Νταλή και να διασφαλίσω κάποια συνέχεια στο έργο του η Όλαφ από τη δικιά της την πλευρά έχει τα δικά της επιχειρήματα και το δικό της έργο. Δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Τώρα με ρωτάτε για τα τρόφιμα. Φυσικά θα είναι σε θελοντική βάση ή το να ενημερώνεται κάποιο. Αλλιώ θα επιβάλαμε μαθήματα για τα πάντα. Πάει να παντρευτεί κανεί, να του κάνουμε ένα μάθημα. Θα φάει να του κάνουμε μάθημα κτλ. Λοιπόν, εγώ ε, δεν πιστεύω ότι θα πούμε στον κόσμο αυτό πρέπει να το τρώτε, αυτό δεν πρέπει να το τρώτε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο πρώτον για τα συστατικά των τροφίμων και δεύτερον για τις επιπτώσεις που έχουν ε, αυτά. Έτσι κι αλλιώς είμαστε ανοιχτοί στην ε, καινοτομία Είμαστε ανοιχτοί και στα εναλλακτικά φάρμακα, εφόσον βέβαια είναι ασφαλή. Από εκεί και πέρα εμείς δεν πρέπει να πειράζουμε τον καταναλωτή, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να επιλέξει το φάρμακο το οποίο προτιμάει. γιατί εδώ παίζουν ρόλο και ψυχολογικοί παράγοντες και μπορεί να προτιμήσει κάτι το οποίο τον ανακουφίζει. Σίγουρα υπάρχει το θέμα των αναλλακτικών φαρμάκων μελετάμε, ετοιμάζουμε και μια έκθεση για το θέμα της διαθεσιμότητας των φαρμάκων, είτε είναι νέα, είτε παλιά, είτε παραδοσιακά, είτε εναλλακτικά. Συνεπώς, για το θέμα αυτό δίνουμε προτεραιότητα στην ελευθερία του πολίτη να επιλέξει, εφόσον βέβαια διασφαλίζουμε ότι ένα φάρμακο είναι σίγουρο και δεν κάνει κακό. Ό,τι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται γίνονται για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία. Αλλά εδώ σταματάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Δεν σας επιτρέπω συμπληρωματική γιατί σας είπα ότι ήταν εκτός θέματος της Επιτροπής μας οι ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Το λόγο... Δία του ευχαριστώ σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε πολλά ζητήματα όπως την ασφάλεια των προϊόντων, το βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που εσείς σκοπεύετε να προτείνετε στους καταναλωτές. Πρόεδρε, εδώ ήθελα να σταθώ σε ένα πρόβλημα που είναι ε, κρίσιμη σημασία για όλου και μάλιστα και όλου του επιτρόπου ασχέτω χαρτοφυλακίου. Κάτι που αφορά του πάντε. Κύριε ε, υποψήφια επίτροπε, ξέρετε ότι θα εκπροσωπήσετε 500 εκατομμύρια καταναλωτέ. Ποια άποψη έχετε εδώ για το άρθρο 21 ε, που εσεί ο ίδιο αναφέρατε. Αισθάνομαι υποχρεωμένη να το αναφέρω αυτό, διότι τοποθετηθήκατε για την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, για τα ζεύγη δύο φύλου. Ποια είναι η δράση που αναλάβετε κατά της ε, διακριτικής μεταχείρισης και των διακριτικών μεταχειρήσεων. Κύριε Μπόρκ. Η απάντηση είναι ναι, όχι γιατί υπάρχει εσωτερική αγορά, αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό. Το άρθρο 21 περιλαμβάνεται στην χάρτα μα. Κάτι κατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή και στη Μαλτέζικη νομοθεσία το άρθρο 21. Είναι κάτι που έχει γραφεί στην πέτρα της νομοθεσίας μας, για να το πω έτσι, Το έχει χαρακτήσει στο μάρμαρο της νομοθεσίας για το σεβασμό της γυναίκας και του σχέσεων ιδίου φίλου στη Μάλτα. Αφού το στηρίζω στη δική μου τη χώρα, γιατί να με το υποστηρίξω και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε την ε, διασφάλισή μου για το θέμα αυτό. Τη δέσμευσή μου. Και γιατί αυτό ήδη συμβαίνει, γιατί άσχετα με το άρθρο 21, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι στη χώρα του τα πάντα πάνε ε, σύμφωνα με το άρθρο 21 και όλα είναι αρμονικά και υπέροχα. Όχι, το άρθρο 21 δεν περιορίζεται στην υγεία, στην ελευθερία, αλλά σε όλε τι υποσχέσει τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν διαφωνώ ελαφρώς με το ποιες είναι πρωτοβουλίες νέες ή όχι για τον καταναλωτή. Έχουμε το ADR που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαπραγματεύσεις, το ODR, επίσης το πρόγραμμα για τους καταναλωτές, με συγκεκριμένες δράσεις εντός του προγράμματος αυτού. Η πρόταση οδηγίες για την πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς επίσης ετοιμάζεται. Επίσης για την ασφάλεια των προϊόντων υπάρχει οδηγία, ε, πρόταση οδηγίας μάλλον, νομίζω σε συνεργασία με άλλους επιτρόπους μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο κ. Σταγιάννη. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, αλλά θέλω να επικεντρωθώ σε λιγότερες που θα θεωρώ ότι μάλλον θα πετύχουν, παρά να τρέξω πίσω από σωρία πρωτοβουλειών και καμία να μην οδηγηθεί σε αίσιο Όχι, εγώ πιστεύω στην στόχευση. Εάν με εγκρίνεται, εάν διοριστώ, Στη θητεία αυτή θα έχω περιορισμένο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μου. Βεβαίω θα ασκήσω τα καθήκοντα μου όπω οι υπόλοιποι επιτρόποι, αλλά μόνο για 10 μήνε. Βεβαίω, κανένα επίτροπο δεν μπορεί να σκέφτεται την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να θέσει ήδη τα θεμέλια για τη μελλοντική του σταδιοδρομία. Σίγουρα. Όμω θέλω να επικεντρωθώ σε κάποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε και σα υπόσχομαι αυτέ που θα αναλάβω να τι φέρω πέρα. Ευχαριστούμε, κυρία Τρούνεν. Συμπλήρωση. Σα ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Για τι ε, συλλογικέ διαφορών έχει γίνει πολλή λόγο. Συγγνώμη, ε, συμπληρώσω πρώτη σα ερώτηση υπάρχει συσχετισμό, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ακόμη για, τον, για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Νέε πρωτοβουλίε θα υπάρξουν, θα συμπληρώσετε τα θέματα δικαιώματων και συλλογική επίλυση διαφορών για του καταναλωτέ. Και θα επιστρέψω στο άρθρο 21. Ενεργός υποστήριξη δηλαδή του πλαισίου LGBT όπως έχει πει και η κυρία Ρέντιν και έπειτα θα στηρίξετε ε, ενεργά το υποσυζήτηση έργο και τη σχετική χρηματοδότηση για την αναπαραγωγική, αναπαραγωγική υγεία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Εάν υπάρξει πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ, που είναι συνυπεύθυνη για τέτοια δικαιώματα, δεν υπάρχει κανένα λόγο να, μην, κανένας λόγος να μην υποστηρίξω τέτοια προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 21 και την ίδια τη χάρτα. Για το πρόγραμμα αυτό που είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου Ανάπτυξης έχω ήδη απαντήσει. Δεν θα παραλείψω να κάνω τίποτε που προβλέπετε. Ούτε θα αφαιρέσω κάτι από το πρόγραμμα, δεδομένου ότι το πρόγραμμα συνάδει με τις νομοθεσίες των ίδιων ε, των κρατών μελών. Τώρα για τη συλλογική διθέτηση τύφρων. με ρωτήσετε ποια είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι σαφή η προσωπική μου τοποθέτηση. Είμαι υπέρ των συλλογικών αντικών μέσων, τη συλλογική ε, διαθέτηση διαφορών και ψήφισα και στο Κοινοβούλιο πέρσι το καλοκαίρι, νομίζω, για την εισαγωγή για πρώτη φορά στη Μάλτα τέτοια νομοθεσία που να προβλέπει τη συλλογική διαθέτηση διαφορών. Βλέποντα τα στατιστικά στοιχεία, νομίζω 18 από τα 27 κράτη-μέλη ήδη έχουν εγκρίνει τέτοια νομοθεσία. Πρόεδρε, παρακαλώ λάβετε υπόψη σα ότι κάθε σχετική οδηγία χρειάζεται να είναι καρπό συνεργασία ε, κι άλλων επιτρόπων με μένα. Θα ήταν λοιπόν αρκετά υπεροπτικό από μέρου μου να πω ότι θα ακολουθήσω τη μια την άλλη γραμμή. Όχι. Αλλά σίγουρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίε. Και ήρθε η ώρα κάποιο βήμα προόδου να γίνει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Να ζητήσω συγγνώμη Γιατί θα πρέπει να με, να, να με ανεχτείτε λίγο ακόμη ως πρόεδρο. Ο κύριος Μπίλαν. E, Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Η Επιτροπή μας εδώ και καιρό προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση των Ευρωπαίων καταναλωτών προκειμένου αυτοί να μπορούν να διαλέξουν τα προϊόντα που θέλουν και να είναι προστατευμένοι. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. Εσείς έχετε εμπειρία από το Κοινοβούλιο της χώρας σας και ελπίζω ότι η συνεργασία θα είναι πολύ καλή και ότι θα μπορέσετε να στηρίξετε το έργο μας. Θέλω τώρα να ξέρω για την πολιτική καταναλωτών. Τι θα κάνετε για να είναι η πιο σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνετε ώστε το Σώμα των Επιτρόπων να φροντίσει γι' αυτό. Εσείς θα είσαστε ο πρώτος που θα υποστηρίζει τα δικαιώματά τους. Πώς θα γίνει δουλειά λοιπόν στα νομοθετικά, στο νομοθετικό αυτό έργο που καλύπτει και άλλους τομείς. Γιατί υπενθυμίζω ότι είναι μια από τις κύριες προτεραιότητές μας όσον αφορά τη στρατηγική των καταναλωτών. Ο κύριος Μπόρκ. Άρθρο 38 του χάρτη. Λέει ότι οι πολιτικές, οι πολιτικές στο πληθυντικό της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οπότε το θέμα δεν είναι ο κατακαιρματισμός ε, ή ο περιορισμός ε, της προστασίας των ε, καταναλωτών, όλες οι γενικές διευθύνσεις και όλες οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να φροντίσουν ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν να πούμε η προστασία των καταναλωτών είναι ευθύνη της κυρίας Ρέντινγκ ή εφόσον με εγκρίνεται είναι ευθύνη του Μπόργκ. Και οι άλλοι επίτροποι να αγωνούν πλήρως τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών. Όχι, αυτή είναι μια εντολή που έχουμε από τον χάρτη και που πρέπει να εφαρμοστεί απάκρι άκρη. Η ατζέντα μας για τον καταναλωτή έχει να κάνει με την κατάρτιση, την ασφάλεια, την ενημέρωση, αλλά επίσης και την επιβολή και την επίλυση, εφόσον υπάρχουν διαφορές. Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ εδώ πολύ, αλλά το κλειδί των Πάντων, εγώ τις είπα αυτές τις τέσσερις αρχές, αλλά το κλειδί βρίσκεται στην ίδια την επίλυση. Γιατί είναι περιττό να έχουμε δικαιώματα και μετά να μην υπάρχει τρόπος γρήγορης επίλυσης εφόσον δεν υπάρχει εφαρμογή. Συνεπώς για μένα υπάρχουν αυτές οι αρχές, υπάρχει η επίλυση, πολύ βασικό, και θέλω να διασφαλίσω ότι η προστασία των καταναλωτών βρίσκεται παντού σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή απάντηση. Κύριε Μπίλαν, έχετε συμπληρωματική, ε? Ναι. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της ενημέρωσης και της κατάρτισης, της διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών. Από τα μέσα που υπάρχουν για να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών, είτε το ECCNet, είτε άλλα κέντρα, είναι συστήματα που πιστεύετε ότι φτάνουν, είναι αρκετά υψηλού επίπεδου και αν όχι, τι θα έπρεπε να κάνετε για να πετύχουμε βελτίωση των μηχανισμών αυτών των ήδη υπαρχόντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρκ. Φυσικά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, αλλιώς δεν θα είχα λόγο εδώ ως Επίτροπος. Πιστεύω όμως ότι έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία που πρέπει να τα τελειοποιήσουμε. Αναφέρθηκα ήδη στα κέντρα προστασίας των καταναλωτών, τα εθνικά δίκτυα για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθούν σε μια εσωτερική αγορά των 500 εκατομμυρίων. Αναφέρθηκα στο βαθμολόγιο, αλλά υπάρχουν και μελέτες. Μερικές φορές ε, οι μελέτες κοστίζουν πολλά, δεν αποδίδουν αρκετά, αλλά υπάρχει μία που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των καταναλωτών και που μας ενδιαφέρει άμεσα γιατί μιλάει για την απογοήτευση των καταναλωτών από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και χάρη στην μελέτη αυτή για τη συμπεριφορά των καταναλωτών εκδόθηκε οδηγία για τα tick boxes, δηλαδή όταν αγοράσει κανείς ένα προϊόν ε, μέσω του διαδικτύου, χωρίς καν να το καταλάβει και χωρίς καν να έχει βάλει σταυρό σε κάποιο τετραγωνάκι, υπάρχει ήδη από πριν αυτό σταυρό στο τετραγωνάκι και είναι σαν να έχει ήδη εγκρίνει κάποια πράγματα. Αυτό απορρέει από μία μελέτη που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες μας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και που έδωσε πραγματικά αποτελέσματα. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ακόμα τέτοιου είδους εργαλεία. Θα συνεχίσω. Ευχαριστώ. Δεν είστε τώρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μπόρχ. Δυστυχώς, δεν έχουμε απαλλαγή από τις διακρίσεις ούτε στο θέμα των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών. Μερικές φορές πάει ένα ζευγάρι σε κάποιο ξενοδοχείο, τους αναγκάζουν να πάρουν δύο δωμάτια αντί για ένα. Λοιπόν, υπάρχουν διακρίσεις ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εσείς που είσαστε, θα είσαστε επίτροπος αρμόδιος για τους καταναλωτές, θα φροντίσετε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε σχετικές οδηγίες και να φροντίσετε να γίνει το σωστό lobbying στις χώρες μέλη ώστε να εφαρμόσετε την οδηγία. Κάτι ακόμα. Πώς εσείς ε, ορίζετε το θέμα του αγώνα για τα δικαιώματα των καταναλωτών εφόσον είσαστε θα είσαστε αρμόδιος για τέτοια θέματα επίτροπος. Ο κύριος Μπόρχ. Κοιτάξτε, προς το παρόν είμαι βουλευτής στην Μάλτα και συμμετέχω και σε διάφορους ομίλους στη Μάλτα. Ελπίζω ότι αυτό δεν πλήττει ε, τη δουλειά μου. Δεν συμμετέχω σε εμπορικές δραστηριότητες. Παλιότερα ναι, αλλά δεν είμαι πια ε, διευθυντής κάποιες επιχείρησης, ούτε έχω τέτοιου είδους οικονομικά συμφέροντα. Από τη στιγμή που έγινα υπουργός, εγκατέλειψα πλήρως και το δικηγορικό μου γραφείο. Οπότε ούτε με αυτό έχω καμιά σχέση, δεν πληρώνομαι από εκεί. Έχω εγκαταλείψει βασικά τους πελάτες μου. Εντάξει, ήμουν υπουργό δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Δεν θα έπρεπε να είχα την παραμικρή σχέση με το δικηγορικό μου γραφείο. Αν κάποιο το έβρισκε αυτό, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Τώρα έχω ήδη απαντήσει για το άρθρο 21. Τι κάνουμε. Το βάζουμε στο κάδρο και το κρεμάμε. Όχι. Πρέπει να το εφαρμόσουμε. Να το εφαρμόσουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Και σας έχω ήδη αναφέρει κάποιο. Έχει να κάνει με την ε, αιμοδοσία, αλλά όχι μόνο. Στη Μάλτα υπάρχει νέα νομοθεσία που έφτιαξα μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οποιοδήποτε νοσοκομείο μπορεί να θεωρήσει τον ε, σύντροφο σαν ε, αρμόδιο για να δώσει την άδεια για κάποια εγχείρηση, για κάτι άλλο που πρέπει να συμβεί στον σύντροφό του. Είπα και πριν ότι υπάρχουν θύλακες διακρίσεων. Αυτό ισχύει. Στο βασιτό άρθρο 21 θα φροντίσω να γίνουν οι αλλαγές που επιβάλλονται για να μην υπάρχουν πια αυτοί οι θύλακες ανισοτήτων. Ο κύριος ευχαριστώ. Μόλις μου έδωσε ο κύριος Γκρότε επιστολή του κυρίου Λένε που λέει ότι έχει εξετάσει η νομική επιτροπή την δήλωση συμφερόντων του κυρίου Μπόρκ και φαίνεται πως υπάρχει κάποιο λάθος Εκτός από αυτό, δηλαδή κάποιο τυπογραφικό σφάλμα, εκτός από αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μπορεί να του προσάψει η Νομική Επιτροπή. Τώρα, είσαστε μέλος σε ορισμένες λέσχες. Δεν κατάλαβα πολύ καλά, είπατε band clubs, band clubs. Εννοώ δηλαδή φανφάρες, ορχήστρες. Κάθε χωριό στην πατρίδα μου έχει και μια ορχήστρα, μια λέσχη ορχήστρας. Και είμαι επίτιμο μέλος ορισμένων τέτοιων, ε, βέβαια, κατά σύμπτωση βρίσκονται στην εκλογική μου περιφέρεια. Δεν θα ρωτήσουμε τι όργανο παίζετε εσείς. Ντένις, νομίζω έχετε ακόμα μια συμπληρωματική ερώτηση. Αν μπορείτε, παρακαλώ, την κάνετε με τρόπο σύντομο. Ευχαριστώ, ναι, για τις αρμοδιότητές σας. Δεν άκουσα τίποτα και θα ήθελα να μου το ξεκαθαρίσετε αυτό. τι θα κάνετε εφόσον υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που οδηγούν σε διακρίσεις στις χώρες μέλη. Πέρα από το άρθρο 29, εσείς τι θα κάνετε όταν διαπιστώνετε τέτοιου είδους διακρίσεις. Ναι, ούτε και αυτό τεχνικά είναι δικιά μας αρμοδιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει αν θέλει ο κύριος Μπόρκ θα απαντήσει. Ναι, σε όλη την πολιτική μου ζωή και την νομική μου καριέρα έχω καταπολεμήσει τις διακρίσεις, οπότε δεν βλέπω γιατί να μην το κάνω αυτό τώρα. Σας ανέφερα ήδη κάποιες πρωτοβουλίες που ανέλαβα ως δικηγόρος, ως υπουργό για να καταπολεμήσω τις διακρίσεις που υπήρχαν και έπαψαν σε ορισμένες περιπτώσεις το κατάφερα αυτό γιατί εγώ πιστεύω στην αξιοπρέπεια του ατόμου και δεν θα πρέπει να υπάρχει τη διάκριση. Κάποιες διακρίσεις είναι αποδεκτές. Αν, ας πούμε, μπορέσω να παρκάρω στο κοινοβούλιο εγώ, φαντάζομαι ότι εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος, αυτή η διάκριση αιτιολογείται. Αλλά γι' αυτό λέω ότι βασίζομαι στον χάρτη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταπολεμώ τις διακρίσεις. Είμαι ξεκάθαρος αυτό γιατί πιστεύω στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία τώρα μακρά ερώτηση ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Πολλές ευχές για επιτυχία. Γιατί εγώ θαυμάζω την νήσο από την οποία προέρχεστε, την οποία θεωρώ μια νήσο ελευθερίας. Και δίκιο έχετε να είστε υπερήφανος. Τώρα, για μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέγεται ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί το ελεύθερο εμπόριο προϊόντων που δεν έχουν την ετικέτα ΨΕ. Όμως δεν ε, είναι προς ε, συμφέρον των καταναλωτών να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν. Βεβαίως το Made in είναι άλλο θέμα αλλά δεν συμφωνείτε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει για το θέμα αυτό του made in ή θεωρείτε ότι δεν είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής. Ακόμη και για στοιχεία γεωγραφικά, γεωγραφικά και οικονομικά ταυτόχρονα προέλευσης. Στη χώρα μου υπάρχει θέμα και με φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και παιχνίδια που προέρχονται από χώρες που δεν χρειάζεται να κατονομάσουμε για να ξέρουμε ποιες είναι, αλλά εννοούμε την Κίνα και που τέλος πάντων μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Η διαφάνεια και ολοκληρώνω. Η διαφάνεια του επιγραμμικού λοιπόν εμπορίου είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. Κύριε Μπορκ, κύριε Μποργέτσιο, συμφωνώ μαζί σας. Έχετε δίκιο στη διαπίστωση ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των προϊόντων αυτών που εισάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν έχουμε το ίδιο σύστημα ελέγχου που έχουμε λόγω χάρη για τα τρόφιμα. Τρόφιμα που εισάγονται και αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κίνδυνος βεβαίως, ο κίνδυνος παραμένει. Διότι ακόμη και αν πρόκειται για μη γεωργικά προϊόντα, για προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, εισάγονται παρόλα αυτά σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον κίνδυνο. Υπάρχει ενδεχόμενο κίνδυνο για τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών. Δεν μπορώ να δώσω υπερβολικά πολλέ λεπτομέρειε, διότι γνωρίζω καλά το θέμα αυτό του, e, του σήματο αυτού αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βεβαιωθώ ότι η ασφάλεια θα αποτελέσει προτεραιότητα. Και για μένα και για όλη την Επιτροπή. Και ίσως έτσι να προχωρήσουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε δηλαδή και για την ασφάλεια των υπηρεσιών. Των υπηρεσιών που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαρκώ μιλάμε για εμπορεύματα και προϊόντα, αλλά όχι για υπηρεσίε ή η ασφάλεια κατά της πυρκαγιάς. Κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις πυρκαγιές γιατί ξέρουμε πόσα θύματα μπορούμε να προλάβουμε έτσι με τα απαραίτητα μέτρα. Θα με απασχολήσει λοιπόν η πράσινη δίπλος για να αρχίσει και ένας γύρος διαβουλεύσεων. Θα δούμε, αλλά Θέλω να έχω την ενεργό συμμετοχή και των υπολείπων συναδέλφων στο κολέγιο. Κάτι που να ξεπερνά αυτά που τώρα αναφέρεται. Υπηρεσίες και ασφάλεια υπηρεσιών στο διαδίκτυο ας πούμε. Ένα, μια εσωτερική αγορά ασφαλέστερη, όπως και εσείς το επιθυμείτε. Κύριε Μποργέτσιο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ συνοπτικά για το εμπόριο στο διαδίκτυο και τα σχετικά παίγνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έλαβε γνώση και τεκμηριωμένη μάλιστα γνώση από ειδικού για την επικίνδυνη δράση εγκληματικών και μαφιόζικων οργανώσεων σε αυτόν τον τομέα. Δεν πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην προστασία των καταναλωτών όχι μόνο από το οργανωμένο έγκλημα αλλά και από τους καταναλωτές που είναι εκτεθειμένοι στα στοιχήματα. Καταλαβαίνετε τι είδου ε, προϊόντα μπορούν να προωθήσουν πρακτορία που όλοι αυτοί οι ευγενείς διαχειρίζονται. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας. Για τον επιπλέον λόγο ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα αγαθό. Είναι κάτι δίκαιο και σωστό. Όμως είναι σαν ένα μαχαίρι που μπορεί να είναι δίκοπο. Δηλαδή μπορεί και καλό να κάνει, αλλά και να δώσει το έναυσμα σε εγκληματικές οργανώσεις που δεν έχουν ευγενείς προθέσεις, να χρησιμοποιήσουν την εσωτερική αγορά όπως χρησιμοποιούν και το χώρο Σέγγεν για να ασκήσουν ή να παραβιάσουν δικαιώματα που τα έχουμε παράσχει στους καταναλωτές μας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με αυτό, διότι υπάρχει σχετική οδηγία, όμως δεν είμαι βέβαιος ότι η υλοποίηση ε, είναι ιδέουσα. Θα αποτελέσει λοιπόν προτεραιότητά μου να ασχοληθώ με το θέμα αυτό στα πλαίσια της θητείας μου. Ελπίζω να έχω τη χαρά βέβαια να με εγκρίνετε για το σκοπό αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Τρεις τώρα βραχίες ερωτήσεις, 50 δευτερόλεπτα αναερώτηση και 2 λεπτά ανααπάντηση. Πρώτος, Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον Αύγουστο υπέβαλα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Brain Packaging για τις brand packaging, για τσιγάρα δηλαδή, οποίο η συσκευασία δεν φέρει φίρμα, δεν φέρει εμπορική ονομασία. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση ήδη το 2012. Ερώτηση. Έχετε κάποια ενημέρωση για το καθεστώς, για την φάση στην οποία βρίσκεται αυτή η πρόταση, διότι εν τέλει διακυβεύονται χιλιάδες θέσεις εργασίας στη σχετική βιομηχανία. Τέλος, η ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτές τις ε, συσκευασίες πειρατεία, λαθρεμπόριο και τέλος άρθρο 17, 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ποια είναι η θέση σας επίσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μείωσης της κατανάλωσης καπνού. Ποια είναι η διασύνδεση με αυτά, με αυτά τα πακέτα τα οποία δεν φέρουν καμιά επωνυμία είναι δύσκολη, να, δύσκολη στην απάντησή της ερώτηση αυτή, διότι η οδηγία ακόμα καλύπτεται από εμπιστευτικότητα. Μπορώ να σας δώσω λοιπόν την προσωπική μου, καθαρά προσωπική μου άποψη, δεν δεσμεύω με κανένα τρόπο εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδα αυτές τις σκέτες συσκευασίες και θα μπορούσαν όντως να είναι αποτελεσματικές. Δηλαδή η οδηγία. Αν τώρα έχουμε φτάσει στην φάση που να μπορούμε να υποχρεώσουμε στην συμπερίληψη στην οδηγία αυτό του plain packaging δεν το ξέρω. Κάτι όμως θα πρέπει να περιλαμβάνεται πάνω στη συσκευασία. Είπα ήδη ότι τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να έχουν και τη μορφή προϊόντων καπνού και όχι κάποιο άλλο πράγματος. Και θα πρέπει και να έχουν τη γεύση προϊόντων καπνού. Αυτή, είναι ο γενικός προσανατολισμός όπου θα πήγαινα εγώ. Αυτό είναι σαφές και εδώ δεν ε, αποκαλύπτω οποιασδήποτε διατάξεις της οδηγίας. Ενδέχεται ορισμένε λεπτομέρειε ήδη να έχουν διαρρεύσει. Εγώ δεν πρόκειται να τη σχολιάσω, δεν πρόκειται να τη σχολιάσω δηλαδή καν την ίδια την οδηγία. Η μόνη χώρα η οποία ήδη έχει περιλάβει νομοθετικέ διατάξει για το plain packaging είναι η Αυστραλία. Έχω δει ορισμένα πακέτα τα οποία καθιστούν λιγότερο ελκυστική την αγορά των προϊόντων αυτού Έγινε προσφυγή στο ανώτατο αυτολληνικό δικαστήριο και στις 15 Αυγούστου απερίφθη η προσφυγή αυτή. Τώρα βεβαίως έχουν προσφύγει ήδη στον ΠΟΕ και υπάρχουν και άλλες περιπλοκές. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε τις χώρες μέλη ελεύθερες ώστε ατομικά, εάν επιθυμούν, να εισαγάγουν τις διατάξεις για το plain packaging. Όχι όμως να εφαρμοστεί άνωθεν στην φάση τουλάχιστον αυτή. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί το νομοσχέδιο αυτό να υποβληθεί και να ενισχυθεί ή να αποδυναμωθεί. Αλλά δεν θα σχολιάσω περισσότερο την ε, οδηγία περί πρώτων καπνού. Ο κύριος Μπούσουτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπόλτς, σας γνωρίζω και προσωπικά. Όχι μόνο επειδή είμαι στο ίδιο κόμμα με εσά, ε, αλλά και γιατί μένω τρει δρόμου πιο κάτω από εσά. Και βεβαίω έχουμε και μια ορχήστρα εκεί. Πάντοτε σα θαύμαζα για την ακαιρεότητά σα, αλλά και διότι στη χώρα μα είστε σύμβολο τη δημοκρατία και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που όλοι ασπαζόμαστε εδώ. Και σας ευχαριστώ, διότι χωρίς ανθρώπους όπως εσείς η χώρα μας, η χώρα μου, δεν θα ασπαζόταν τις ευρωπαϊκές αυτές αξίες. Ερώτηση τώρα. Πώς εσείς ως Επίτροπος θα προστατεύσετε τους καταναλωτές από τις παραπλανητικές πρακτικές. Για παράδειγμα, επιθετικέ πρακτικές από επιχειρήσεις οι οποίες εξαπατούν καταναλωτές και τους οθούν να αγοράσουν εμπορεύματα τα οποία ποτέ δεν θα αγόραζαν. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε το φαινόμενο αυτό. Κύριε Μπούσουτιλ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Προσθέτω ότι αυτό που αναφέρατε, ιδιαίτερα, το έβλεπα προπολών ετών στη δικηγορική μου πρακτική μεταξύ 1980 και 1995, όταν ερχόντουσαν στο δικηγορικό μου γραφείο κάποιοι με ένα λογαριασμό στα χέρια τους και εμφανιζόταν τελικά να έχουν παραγγείλει κάτι το οποίο διόλου δεν είχαν θελήσει, κυρίως οι κυκλοπαίδειες τότε και δεν υπήρχαν καν τα online, τα επιγραμμικά τότε. Εγώ δεν αγοράζω βιβλία online, πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο, αλλά όλο και περισσότεροι άνθρωποι ας πούμε οργανώνουν διακοπές τους επιγραμμικά. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις, είτε πρόκειται για τα λεγόμενα directories, είτε ακόμα και φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία πολλούνται καμιά φορά επιγραμμικά. Αν δεν εξετάσουμε πραγματικά τι συμβαίνει στι διάφορε χώρε μέλη, θα καθυστερούμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και δεν θα ανταποκριθούμε στι υποχρεώσει που έχουμε απέναντι στου καταναλωτέ. Μίλησα ήδη για τα εργαλεία που έχουμε, αποζημίωση ODR, ADR, τα διάφορα βαθμολόγια, scoreboard, τα κέντρα προστασία καταναλωτών, αλλά και να εξετάσουμε και την έκθεση που πρόκειται να υποβληθεί για το τι γίνεται επιγραμμικά. Και αυτά που συμβαίνουν δεν είναι πάντοτε ευχάριστα. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σε εγρήγορση. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι ιδιαίτερα άγρυπνος φρουρός και όπως και για τους ισχυρισμούς υγείας που αφαιρέσαμε την βάση, το ίδιο πρέπει να κάνουμε για τέτοιες πρακτικές στο εμπόριο online. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών. Ευχαριστώ. Πρέπει ε, να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά κύριε Πόργο, εσείς πώς θα εφαρμόσετε ένα συνολικό πακέτο για τα δικαιώματα του καταναλωτή όταν ξέρουμε ότι το χαρτοφυλάκιό σας ουσιαστικά είναι μοιρασμένο μεταξύ διαφόρων επιτρόπων το οποίο κάνει την κατάσταση κάθε φορά πολύ δύσκολη. Για παράδειγμα αυτά που ανέφερε και ο συνάδελφος για τις ε, συλλογικές ε, προσφυγές. Πρόσφατα προτάθηκε ένα νομοθετικό πακέτο για τα δημοσιονομικά μέσα. Εσείς τελικά τι μέσα θα εφαρμόσετε ώστε να διασφαλίσετε ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να προστατευτούν συλλογικά μέσω αυτών των εργαλείων. Τώρα έρχομαι στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αντιλαμβάνομαι καλά αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή δεν θα έχετε καμία επιφύλαξη στο έργο σας. Θα απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα γιατί βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν θα έδειχνα αρκετό πατριωτισμό αλλιώς. Συνεπώς, σας ευχαριστώ βέβαια για την ερώτησή σας και ξέρω πολύ καλά πόσο δραστήριος είσαστε γιατί έχω ενημερωθεί κι εγώ. Σίγουρα η αν εγκριθεί αυτό το θέμα θα κάνει κάποια διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υπέρ βέβαια των συλλογικών προσφυγών και των συλλογικών επιλύσεων και είναι κάτι το οποίο το έχω συζητήσει και με άλλους επιτρόπους. Εσείς λέτε ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι μοιρασμένο, είναι αρμοδιότητα δηλαδή πολλών επιτρόπων συγχρόνως. Εγώ όμως θα είμαι επίτροπος και γι' αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω αυτήν την ε, παρατήρηση. Κάτι αντίστοιχο είχατε ρωτήσει και το προκάτοχό μου και είχε απαντήσει. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τις αρμοδιότητες που έχει η κυρία Ρέντινγκ, η οποία ασχολείται και αυτή με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συνεπώς, ο ρόλος μας είναι να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές ιδιαίτερα για τα θέματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών. Με ρωτάτε επίσης κατά πόσο θα είμαι πλήρως, θα συμμορφωθώ πλήρως με τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων χωρίς επιφυλάξεις. Εγώ έχω μελετήσει το χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων και δεν βλέπω τίποτα που να με εμποδίζει. πρέπει να δούμε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν έχω επιφυλάξεις λοιπόν όσον αφορά τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καμία επιφύλαξη. Και μπορώ να πω ότι ο χάρτης ο ίδιος δεν προβλέπει εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις. Κάθε δικαίωμα λοιπόν που προβλέπεται τελειώνει στα σύνορά μας. Αλλιώς δεν υπάρχουν επιφυλέξεις, το λέω και επιμένω σε αυτό και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Πάντα στη ζωή μου αγωνιζόμουν κατά των διακρίσεων. Όλοι βέβαια κάνουν κάποια σφάλματα στη ζωή τους, αλλά πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτά είναι πράγματα τα οποία υποστηρίζω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και για μένα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς όλους σας για τις ερωτήσεις μέχρι τώρα και τώρα ο κύριος Γκρόντε πάλι έχει το λόγο, να αναλαμβάνει την Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Ερχόμαστε τώρα στον τέταρτο γύρο. Και τώρα πια την σκητάλη παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Γεωργίας. Πρόκειται λοιπόν για πέντε βραχίες ερωτήσεις, των 50 δευτερολέπτων δηλαδή για τον ερωτώντα και δύο λεπτών για την απάντηση από τον κύριο Μπόργκ. Πρώτος, ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπόρκ, απλή ερώτηση. Το Ευρωκοινοβούλιο στις 18 Δεκάτου 2010 έλαβε την εξής απόφαση ζήτησε οι αγροτικές εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνονται, να επιτρέπονται μόνο εφόσον για τις εισαγωγές αυτές ισχύουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές προστασίας καταναλωτού, φύσεως και ζώων και ταυτόχρονα κοινωνικά ελάχιστα στάνταρτ. Πρόκειται για ε, απόφαση που ελήφθη με πλειοψηφία 535 ψήφων. Θα τη σεβαστείτε? Ευχαριστώ κύριε Μπόλ και εσείς. Α, βεβαίω. Πολλά μπορώ να σα απαντήσω. Κοιτάξτε, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Θα ήταν ανέντιμο να κλείσουμε να επιτρέπουμε αφενός εισαγωγές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε ορισμένε ελάχιστε προδιαγραφές και ταυτόχρονα τι ίδιες προδιαγραφές να επιβάλλουμε στους δικούς μας γεωργούς. Είναι βέβαια ευαίσθητο το θέμα και κατανοώ γιατί. Διότι η ενιαία αγορά, αυτή η ελεύθερη αγορά 500 και εκατομμυρίων καταναλωτών δεν θα πρέπει να διακρίνει σε βάρος των ίδιων των Ευρωπαίων αγροτών. Αλλιώς όμως από ότι για την ασφάλεια των προϊόντων που δεν είναι γεωργικά προϊόντα, για τα γεωργικά προϊόντα έχουμε τρόπο να επιβάλλουμε την τήρηση των προδιαγραφών. Έχουμε το FVO, Food and Veterinary Office, που έχει έναν αριθμό επιθεωρητών που επιθεωρούν όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε όλες τις συμφωνίες πηγαίνουν στην Αργεντινή, πηγαίνουν στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες και προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να εξασφαλίσουν ώστε ό,τι εισέρχεται στην αγορά αυτή των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών ανταποκρίνεται στις ίδιες προδιαγραφές που απαιτούμε να εκπληρούν οι δικοί μας αγρότες. Μπορούμε να ενισχύσουμε την επιβολή αυτή. Μπορούμε. Έχουμε και τη δέσμη μέτρων για ε, μέτρα ελέγχου για την προστασία της υγείας ε, ανθρώπων, ζώων και φυτών και έχουμε βέβαια και τις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες. Γνωρίζω ότι και η Ρωσία εντάχθηκε στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπόριου. Υπάρχουν βέβαια κάποια αμφιλεγόμενα θέματα σχετικά με το τι εισάγεται και με το τι δεν επιτρέπεται τρέπεται να εξαχθεί από εμά προς αυτούς για τεχνικού λόγους, δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες αυτούς για λόγους προστατευτισμού, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μένουμε ώστε και οι άλλες χώρες να τηρούν τις υποχρεώσει που έχουν αναλάβει με την είσοδό του στον ΠΟΕ. Και σας βεβαιώ ότι θα επιμείνω στην ανάληψη αυτών των υποχρεώσεων. Λούις Κάπολα Σάντος, 50 Ευχαριστώ Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, πριν από μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε να αντιμετωπίσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η ασθένεια, η νόσο των τρελών αγελάδων. Θυμόμαστε ότι για να εκριζωθεί το πρόβλημα αυτό λύθησαν ε, ριζικά μέτρα καταστρέφονταν ε, και το κρέας και τα κόκαλα των ζώων που σφαγιάζονταν. Και βεβαίως θυμόμαστε πόσο μεγάλο θέμα υπήρχε με όλα τα μερικαστικά. Ε, αργότερα υπήρξε και απαγόρευση για την ε, χρήση των υλικών αυτών στις ζωοτροφές. Γιατί υπήρχε κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης και ρήπανσης στο επίπεδο μετάδοσης μάλλον στο επίπεδο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. και λοιπόν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται συστηματικά οι καταναλωτέ προκειμένου να διαλυθούν και να διασκεδαστούν αυτέ οι επιβολίε. Κύριε Επίτροπε, τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα αυτό, εφόσον αναλάβετε τα καθήκοντά σα και ευθύ εξ αρχή. Κύριε Μπόρκ, το πρόβλημα αυτό το γνωρίζω κάπω. Διότι όταν υπήρξε η νόσος, ε, τους πογκόντους κεφαλοπάθειας και σχετικό, τα σχετικά κρούσματα, γνωρίζω τι συνέβη, διότι ακριβώ υπήρξαν τεράστιες οικονομικές συνέπειες στις χώρες που επλήγησαν από την ασθένεια. Και κάποιες μάλιστα επλήγησαν με τρόπο οξύτατο. Εκεί ανελήφθησαν σοβαρά μέτρα για να μην χρησιμοποιούνται πλέον πρωτεΐνες, στις ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται για ζώα τα οποία δεν καταναλώνουν κρέας αλλά είναι μυρικαστικά. Σημειώνω ότι υπήρχαν κάποιοι που λένε, έλεγαν και λένε γιατί να μην άρουμε αυτή την απαγόρευση. Τουλάχιστον για τα ζώα που καταναλώνουν κρέας. Εκεί η πρωτεΐνη θα μπορούσε να επιτρέπεται στις ζωοτροφές τους. Όμως, δεν καταλαβαίνω την ε, άρση μιας τέτοιας απαγόρευσης και τον επιτρέπεται η πρωτεΐνη αυτή για τα ζώα τα οποία είναι μυρικαστικά, δεν είναι σαρκοφάγα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε άκρος προσεκτικοί, διότι έχουν περιοριστεί σοβαρότατα τα κρούσματα σποκόδους εγκεφαλοπάθειας μέσα στην παράδοση του χρόνου και χάρη στα μέτρα που υιοθετήσαμε. Και το να γίνουμε επικέστεροι, πιο χαλαροί με την απαγόρευση αυτή, μπορεί να επιτρέψει την ανάδυση μελλοντικών κρουσμάτων. Κανείς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Για μια σειρά λόγων, αλλά και γιατί πρέπει να είμαστε πολύ βέβαιοι και να αισθανόμαστε ασφάλεια για τα δικά μας τρόφιμα. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με άκρα προσοχή εδώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάιον. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Μπόρκ. Η προστασία των ζώων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα μέσα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, ιδιαίτερα η μεταφορά των ζώων. Ο προκάτοχός σας ε, εγκαθίδρυσε έναν διεθνωτικό διάλογο, αλλά δεν στήριξε την πλήρη απαγόρευση Τη μεταφορά πάνω από 8 ώρε όταν τα ζώα πηγαίνουν φαγή. Εσείς ε, τι θέση θα υποστηρίξετε τελικά, θα υποστηρίξετε αυτή τη θέση για την απαγόρευση τη μεταφορά πάνω από 8 ώρο. Ο κύριος Μπόρκ. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεσμεύομαι από τις αποφάσεις της Επιτροπής Μερικές φορές η προστασία των ζώων θεωρείται σαν κάτι το δευτερεύον, σαν κάτι που δεν είναι σημαντικό, σαν κάτι που εμποδίζει την πρόοδο σε μερικούς τομείς. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν βρίσκεται κανείς εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τότε τα επιχειρήματα που ακούγονται είναι «Α, να είμαστε ρεαλιστές», Οπότε, εδώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν θα σας υποσχεθώ κάτι που δεν μπορώ να πετύχω. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ όμως είναι τα εξή δύο. Πρώτον, η τρέχουσα ρύθμιση για την μεταφορά των ζώων Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ακούσει, εγώ δεν έχω ακούσει να υπάρχει παράβαση να υπάρχει καμία διαδικασία, δηλαδή επί παραβάση σε βάρος κάποιας χώρας μέλος, επειδή παραβιάζει τις ρυθμίσεις για την ε, μεταφορά των ζώων. Μιλάω για τις τρέχουσες ρυθμίσεις, έτσι. Βέβαια, πάντα υπάρχει περιθώριο να κάνει κανείς τα πράγματα καλύτερα. Γιατί να μην υπάρχει ένα σύστημα αφού όλα τα οχήματα έχουν γιατί να μην μπορούν να έχουν και αυτά που μεταφέρουν ζώα ώστε να δούνε πώς μπορούν να διευκολύνουν την ε, μεταφορά. Πρέπει επίσης να σας πω ότι υπάρχει μία πρόταση για ένα γενικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία των ζώων και να ξεκινήσει του χρόνου. Ήδη έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Οπότε γιατί να μην ξανανοίξει το θέμα για το κατά πόσο φτάνουν οι σημερινοί κανόνες ή όχι και να δούμε και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμοι ή όχι. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος... Χόισλινγκ. Κύριε Μπόρκ, Είπατε ότι θέλετε η Ευρώπη να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητή για την προστασία των καταναλωτών. Άρα και μηδενική ανοχή ορισμένων εισαγωγών, υποθέτω. Δεύτερο, ασκείται κριτική δικαιολογημένη στην ΕΦΣΑ για αδιαφανείς διαδικασίες και ιδίω για την αξιολόγηση των κινδύνων των GMO, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα ζητήσετε αναθεώρηση των διαδικασιών των ελέγχων αυτών. Και όσο δεν συμβαίνει αυτό και όσο δεν υπάρχει νέα αρρύθμιση και επομένως εδώ κίνδυνος επανεθνικοποίησης των ελέγχων για την εισαγωγή των GMO, θα ζητήσετε ένα μορατόριο για την εισαγωγή τους. Κύριε Μπόλγκ, θα πρέπει να, είμαι, θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για όσα αναφέρονται σε τρόφιμα και άλλο θέμα για όσα αναφέρονται σε ζωοτροφές. Αυτό είναι πολύ αμφισβητήσιμο το αν πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς των μη εγκεκριμένων εισαγωγών. Τώρα, θα στηριχτώ στην ΕΦΣΑ ή όχι. Πρώτα-πρώτα, η ΕΦΣΑ έχει ένα σκοπό που υπάρχει για να προσφέρει δηλαδή πραγματικές ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές. Και σωστό είναι, πάντα είναι σωστό να φροντίζει κανείς ώστε να υλοποιείται αυτή η ανεξαρτησία. Και εγώ θα εργαστώ σκληρά ώστε να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία. Όμως, δεν θα παρατηθώ από τις δικές μου ευθύνες, διότι δεν είναι η ΕΦΣΑ εκείνη η οποία εγκρίνει, αλλά ο Επίτροπος, ο ίδιος ο Επίτροπος. Άρα εδώ εγώ έχω τον τελευταίο λόγο. Δεν θα χρησιμοποιήσω την εύσα για σκοπό άλλο εκτός από το να ζητήσω να μου υποβάλει ξεκάθαρα στέρεα επιστημονικά δεδομένα. Εγώ όμως θα αποφασίσω εάν θα υπάρχει έγκριση γενική ή υπό όρους, είτε υπό όρους έγκριση είτε όροι στην εφαρμογή της έγκρισης. η υπο ειτε υπο εγκριση ειτε όρη στην εφαρμογη της εγκρισης Απάντησή μου λοιπόν είναι ότι όχι δεν θα είμαι δούλος της ΕΦΣΑ, αλλά ούτε θα αγνοήσω τα όσα λέει. Τώρα, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γνωρίζω καλά τις ευαισθησίες του θέματος. Γνωρίζω και το επίμαχον του θέματος. Γνωρίζω πόσο εύκολο είναι για το Συμβούλιο να αφήσει τα πράγματα αυτά στα χέρια της Κομισιόν και να μην προωθήσει η αδίποτε πρόταση, ούτε καν της εφαρμογή της επικουρικότητας σε προτάσεις για καλλιέργεια. Δηλαδή ότι η χώρα, η συγκεκριμένη χώρα, θα είναι ελεύθερη να επιτρέψει την καλλιέργεια ή όχι στην επικρατειά της, εκτός από θέματα βέβαια υγείας και περιβάλλοντος που παραμένουν αρμοδιότητες της Επιτροπής της Κομισιόν. Ευχαριστώ, διακόπτη πρόεδρος. Τελευταίος Νίκολσον, 50 δευτερόλεπτα από τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε, παρόμοιο θέμα. Εμείς στην Ευρώπη χρειαζόμαστε εισαγωγές σπόρων για τις ζωοτροφές μας, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Νότια Αμερική. Για, ποια είναι η θέση σας για τις εισαγωγές τροποποιημένων γενετικά οργανισμών και χρειαζόμαστε άδειε licensing για να αντιμετωπίσουμε και το υψηλό κόστος που αντιμετωπίζει η βιομηχανία σε αυτή την περίοδο. Γνωρίζω τις ευαισθησίες και αυτού του θέματος, απαντά ο υποψήφιο επίτροπος. Και γνωρίζω και όλα τα σχετικά με την επισήμανση του ποσοστού των περιεχομένων ε, ε, GMO που πρέπει να είναι 0,9% και πρέπει να υπάρχουν βεβαίω να πληρούνται ορισμένα επιστημονικά κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την ίδια την καλλιέργεια, γνωρίζω ότι υπάρχει έκθεση Σεραλίνη την οποία θα χρειαστεί να εξετάσω και η οποία εξετάζεται τώρα σε τελική φάση από την ΕΦΣΑ επίσης. Αλλά για τις εισαγωγές θα συμμορφωθώ με τους υφιστάμενους κανόνες, εκτός εάν η ΕΦΣΑ δώσει άλλο μήνυμα. Οπότε τότε θα χρειαστεί να αποφασίσω και να εγκρίνω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εκατομμύρια εκτάρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλλιεργούν μη, γενετικούς, μη ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γνωρίζω τις αντιστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, που το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και θα ήταν ανεύθυνο νομίζω για μένα να μην λάβω υπόψη όλες τις απόψεις και ιδίω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα πέσω λοιπόν με τα μούτρα εκεί όπου χρειάζεται να προπατά κανείς με ιδιαίτερη προσοχή και βεβαίως η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται με εύλογο τρόπο αλλά σε θέματα όπου δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά δεδομένα οφείλει κανείς να καθυστερεί λίγο περισσότερο παρά να προτρέχει. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Υποψήφια, συγγνώμη. Τώρα τελείωσε και ο τέταρτος γύρος. Οι ερωτήσεις των συναδέλφων της Επιτροπής Γεωργίας ολοκληρώθηκαν και οι απαντήσεις δηλαδή και τώρα μπαίνουμε στον τελευταίο γύρο και έχουμε εννέα συναδέλφους οι οποίοι θα θέσουν ερωτήσεις. Πρώτα τρεις μακρές ερωτήσεις Πέντε λεπτά δηλαδή, όπου μπορεί να τεθεί και συμπληρωματική ερώτηση και μετά θα ακολουθήσουν πάλι έξι βραχίες ερωτήσεις. Αρχίζει με μακρά ερώτηση για δεύτερη φορά η κυρία Γιάννα Κουδάκη. Ευχαριστώ. Συζητήσαμε το θέμα του προπολογισμού και χαίρομαι που δεν είσαστε υπερευαίσθητων περικοπών. Αυτό είναι κάτι που τα απαιτούν και οι εκλογέ μα. Ε, Επίση, μιλήσαμε για οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με μεγάλη χαρά άκουσα τι τάσει σα για τη σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ ελπίζω ότι όσα κάνατε στου μουσικούς συλλόγου που δραστηριοποιήσετε δεν θα αντιφάσκουν με τις υποχρεώσεις σα ω Επιτρόπου. Όμω, τι συγκεκριμένα σχέδια έχετε για να συμφιλειώσετε συγκρούσεις συμφερόντων που έχουν να κάνουν με την κακοδιαχείριση την, ε, ε, και την ε, αμφισβητούμενη διαχείριση κονδυλίων από ευρωπαϊκού οργανισμού, όταν προτείνονται ευαίσθητε περικοπέ σε προπολογισμού των οργανισμών αυτών. Ο πρόεδρο κ. Γκρότε. Κύριε Γιάννα Κουδάκη, χαίρομαι που θέτετε δεύτερη ερώτηση, αλλά προσπαθήστε να μείνετε στον τομέα αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρω εάν ο υποψήφιο Επίτροπο επιθυμεί να απαντήσει, διότι δεν είναι θέμα τη ιδιωτικότητά του. Εσεί κύριε Μπόρκ θα αποφασίσετε τι θέλετε τα Πράξτε. Δεν έχει μικρόφωνο, θα. Α, λοιπόν. Είμαι μέλος μουσικού συλλόγου, δεν είμαι ο ίδιος ο ε, μουσικός. Τους υποστηρίζω απλώς. Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να παρεμπληθεί στην, στον χειρισμό από πλευράς μου των ε, φακέλων προστασίας καταναλωτού. Αν υπάρχει έστω και ελάχιστη σχετική παρεμβολή, μην ε, φανταστείτε ότι θα διστάσω έστω και ένα δευτερόλεπτο να παραιτηθώ από τον μουσικό σύλλογο. Τώρα, σύλλογο, για τις εύλογες περικοπές. Το ερώτημα είναι, τι είναι εύλογες περικοπές και σε ποιου τομεί θα πρέπει να επιβληθούν περικοπές, διότι όταν τίθεται θέμα υγείας, εάν περικόψετε με τρόπο αυθαίρετο, Συνήθως οι άνθρωποι υποφέρουν και ιδίω οι πιο ευάλωτοι είτε λόγω ηλικία είτε λόγω περιστάσεων. Υπάρχει τρόπος μείωσης των δαπανών χωρίς απαραίτητα να μειώσετε το επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Έχουμε τα e-health scoreboards, e-health networks, χρησιμοποιούμε δηλαδή ε, συστήματα μακρόθεν ε, παρακολούθηση των ασθενών στο σπίτι τους. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μαθαίνω ότι ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων που προστατεύονται από ευρεσιτεχνία θα γίνουν τώρα γενώσιμα φάρμακα σε λίγα χρόνια, άρα θα μειωθεί το ύψος των δαπανών για τα ίδια τα φάρμακα. Τώρα, οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά τους δύο οργανισμούς που εμπίπτουν στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, δεν είναι τμήμα της ΣΑΝΚΟ, διότι είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί. Αλλά θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις αυτές. Αλλά θα διαβουλευτώ πρώτα με τους άλλους επιτρόπους για να δούμε εάν μπορούμε να θεσπίσουμε κοινού κανόνες για όλους τους οργανισμούς, τους ανεξαρτήτους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μειωθεί ο θόρυβος, διότι είναι πολύ δυσχερής εν τέλει η θέση και του υποψηφίου που επί ένα, επί τρίωρο είναι εδώ μπροστά και απαντά σε ερωτήσεις. Όποιος επιθυμεί να ομιλήσει παρακαλώ να εξέλθει σε αίθουσας. Καρλ Σλούτερ. Ευχαριστώ. Ακούσατε κι εσείς τις ερωτήσεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για τον καπνό, για το αλκοόλ όμως, τι σκοπεύετε να κάνετε. Πιστεύετε ότι πρέπει, γιατί άκουσα τι είπατε, είπατε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Πολλά πράγματα. Υπενθυμίζω όμως ότι στη Μάλτα εσείς Κάνατε πράγματα καταψηφίσατε την δήλωση των Ηνωμένων Εθνών, οπότε θα αλλάξετε τώρα την στάση σας. Πώς εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που θα κάνετε. Ο κύριος Μπόρκ. Στην ε, Μάλτα εγώ δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με το AIDS όπως ε, λέτε. Για το αλκοόλ η δέσμευση είναι σαφής. Υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την καταπολέμηση του AIDS στην γραμμή που σας παρουσίασα, δηλαδή πρόληψη και θεραπεία και ε, πρέπει να φροντίσουμε να απαλείψουμε τον στιγματισμό των ασθενών. Είναι σοβαρό, δεν μπορούμε να παίζουμε με την ανθρώπινη ζωή και με ανθρώπινες τραγωδίες, οπότε είναι σαφής νομίζω η θέση μου. Όσον αφορά τώρα το ενόπνευμα, ξέρω ότι είναι και αυτό κάτι που υπάρχει, όπως υπάρχουν και τα τσιγάρα. Έχω πει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, ασθένειες, αλλά για να τις καταπολεμήσουμε πρέπει πρώτα να καταπολεμήσουμε τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το αλκοόλ. Δεν λέω ότι πρέπει να απαγορευτεί το αλκοόλ, αλλά να εξηγήσουμε τους κινδύνους που απορρέουν από το αλκοόλ στους καταναλωτές, να τους εξηγήσουμε τι μηχανισμοί ε, λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό τους όταν καταναλώνουν αλκοόλ, γιατί μερικές φορές δεν το γνωρίζουν. Και βέβαια το πρόβλημα είναι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συμπληρωματική. Νομίζω ότι δεν είσαστε σαφείς για την ερώτησή μου. Εσείς χρησιμοποίησατε τις δικές σας αρμοδιότητες ως Υπουργός Εξωτερικών στη Μάλτα για να αλλάξετε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά την ε, ε, αναπαραγωγή και την πολιτική τη σχετική στην Ευρώπη. Αυτό είναι για το οποίο σας ρωτάω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όσον αφορά το ΝΟΙΕ. Εγώ ασχολήθηκα με την Μεσόγειο, με την Μέση Ανατολή, με την Μεσογειακή πολιτική, αλλά ως υπουργός Εξωτερικών ποτέ δεν ασχολήθηκα με τα θέματα αυτά γιατί δεν ήταν δικιά μου αρμοδιότητα. Πήγα στην Γενική Συνέλευση τελευταία φορά που ήμουν στα Ηνωμένα ε, Έθνη και αυτό είπα, είπα ότι πήγα εκεί, αλλά εκεί εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό. Δεν πήρα το λόγο. Ασχολήθηκα με πολιτικά θέματα, γιατί αυτή ήταν η αρμοδιότητά μου. Τώρα τα θέματα της υγείας και των καταναλωτών είναι εντελώ διαφορετικά από τις εξωτερικές υποθέσεις. Οπότε αρχίζω να εξοικειώνομαι με τα θέματα αυτά και ζητώ συγγνώμη αν δεν κατάλαβα... Δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα αρκετά καλά κάποιες λεπτομέρειες των θεμάτων αυτών, οπότε αυτό φάνηκε σήμερα στην ακρόασή μου, αλλά ζητώ συγγνώμη, αλλά να ξέρετε ότι τα θέματα για τα οποία δεν είμαι αρμόδιος και δεν ήμουν αρμόδιος δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Η κυρία Λεπάζ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπόργο, θέλω να επανέλθω, επιτρέψτε μου, στο θέμα των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και την πραγματογνωμοσύνη της ΕΦΣΑ. Διευκρινίστε μου το εξή. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση ψήφισε ένα κείμενο για να τροποποιηθεί η οδηγία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Περιμένουμε τη θέση του Συμβουλίου. Εσείς είσαστε υπέρ του να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε δεύτερη ανάγνωση με κείμενο για το οποίο να έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο. Δεύτερον, μας είπατε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ. Καλώς. Σκέφτεστε να υιοθετήσετε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να βελτιωθεί και η εικόνα αλλά και η πραγματικότητα όσον αφορά την ανεξαρτησία του οργανισμού αυτού. Και Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τα συστήματα αξιολόγηση, ιδιαίτερα για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, μια που πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε έχουν ζητήσει τα συστήματα αυτά να τροποποιηθούν. Εσεί θα ξαναδείτε, θα αναθεωρήσετε τι κατευθυντήριε γραμμέ ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρκ. Ναι, είναι σημαντικό η αντίληψη είναι ένα πράγμα, η πραγματικότητα είναι επίσης ε, μια πραγματικότητα όπως θα λέγω ότι είναι και η αντίληψη. Εγώ θα έλεγα ότι τα δύο συνδέονται άμεσα και πρέπει να συνδέονται άμεσα. Δεν ξέρω αν δεν με καταλάβετε καλά, θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Κοιτάξτε κύριε Λαπάζ, εγώ είμαι σαφής για το θέμα της ΕΦΣΑ. Κάθε φορά που η ΕΦΣΑ μας παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα, φυσικά και τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς είπα ότι δεν θέλω να βιαστώ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πάρουμε αποφάσεις. Υπάρχουν συνέπειες και από την ε, μη λήψη απόφασης. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να προσφύγει κανείς ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειψη απόφαση. Θα σας δώσω όμω ένα παράδειγμα. Αν υπάρχει σχετική έκθεση, πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια που θα δοθεί σε μια τέτοια έκθεση. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει αξιολόγηση για την έκθεση αναλύνη είναι σημαντικό να έχουμε μια έκθεση αξιολόγησης από την ΕΦΣΑ πριν προχωρήσουμε σε δράση. Είμαστε συνεπώς σε μια κατάσταση, τη γνωρίζετε, όπου το Συμβούλιο το αφήνει στην Επιτροπή να αποφασίζει. Εξάλλου ο ίδιος ο Επίτροπος δίνει την άδεια και όχι ΕΦΣΑ. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, γιατί αν πάρουμε λάθος αποφάσεις, αυτό προκαλεί ζημιά. Αλλά απόφαση πρέπει να ληφθεί. Ο πρόεδρος Κρότε. Α, ναι, κύριε Λεπάνος, θέλετε συμπληρωματική ερώτηση. Κοιτάξτε, κύριε Μπόρκ, θα απαιτήσετε σε ό,τι αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, μελέτες τοξικότητας μακράς διάρκειας, που δεν υπάρχουν. Δεν κατανόησα καλά όλη την ερώτηση. Με συγχωρείτε. Αν θα, αν θα ζητήσω, θα, θα, θα επαναλάβω, θα επαναλάβω, λέει ρωτώσα. Προτίθεστε να απαιτήσετε μελέτες τοξικότητας μακράς διάρκειας για να γνωρίζετε τις επιπτώσεις στην υγεία των GMO ή θα παραμείνετε μονάχα στις 80 ημέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Κύριε Μπόρκ, σας παρακαλώ. Όπως ξέρετε κυρία Λεπάζ, όταν προσπάθησε η Κομισιόν να επιβάλλει τις 90 ημέρες στις ε, εταιρείε δεν υπήρξε τελικά συμφωνία. Ήδη λοιπόν η αύξηση στις 90 ημέρες προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες, όμως θα βασιστώ στις επιστημονικά δεδομένα. Και βεβαίως θα εφαρμόσω με εύλογο τρόπο την αρχή προφύλαξης. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να επανέλθουμε. Αν αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τα όσα λέει η ΕΦΣΑ για την ε, δοκιμασία 90 ημερών στα ζώα έτσι ώστε να ισχύσει μακροτέρα περίοδος αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βασιστεί σε επιστημονικά δεδομένα. Είμαι βέβαιος ωστόσο ότι η ανεξάρτητη ΕΦΣΑ εφόσον αλλάξει την, ε, ε, ε, συστάσει τη, ε, ω ανεξάρτητη, αυτό θα είναι και το σωστό. Ευχαριστώ. Έξι ακόμα αγορητέ από την Επιτροπή περιβάλλοντο. Άλλοι λοιπόν οι σύντομε ερωτήσει. 50 δευτερόλεπτα η ερώτηση και 2 λεπτά η απάντηση. Πρώτη η κυρία Γιολάντα Χίπνερ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε μέχρι τώρα. Σύντομη ερώτηση. Βρισκόμαστε στην περίοδο εμβολιασμού κατά της γρήπης. Τέτοιες εκστρατείες προβλέπονται και για τα επόμενα χρόνια. Πώς βλέπετε τον ρόλο σας για τη σταθεροποίηση της αγοράς των εμβολίων έτσι ώστε να εγκρίνονται μόνο τα προϊόντα εταιριών τα οποία είναι ασφαλή και δοκιμασμένα. Επίσης, ο πανικός που ξέσπασε πρόσφατα σε σχέση με τους εμβολιασμού. Νομίζετε ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα τέτοιο φαινόμενο και ποια αντίδραση θα έχετε. Κύριε Μπόρκ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εμβολιασμούς. Βεβαίως, πρέπει να αναλύσουμε όλες τις εκθέσεις, τα επιστημονικά δεδομένα, για να διασφαλίσουμε ότι οι εμβολιασμοί θα είναι ασφαλείς. Καμιά φορά πρέπει να αγωνιστούμε και κατά προκαταλήψεων κατά τον εμβολιασμό διότι οι εμβολιασμοί σώζουν ζωές. Κάτι που με ανισχύει ιδιαίτερα όταν υπήρξαν κίνδυνοι για την υγεία στο παρελθόν με το ξέσπασμα επιδημιών, είναι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδράσαμε με ενιαίο τρόπο. Ο καθένας από εμά θεωρήσαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα μόνοι μας. Και όμως και υπό την αρχή της επικουρικότητας, όταν μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα μόνη της, τότε νομίζω ότι η Κομισιόν, το κέντρο, πρέπει να παρέμβουν για να προστατεύσουν τελικά την υγεία των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Και για το ιδιαίτερο θέμα των εμβολιασμών που αναφέρατε, θα πρέπει στην οδηγία για την αντιμετώπιση απειλών υγείας που συζητείται ήδη στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, ε, να συνεχίσουμε μάλλον τη συζήτηση αυτή. Το ερώτημα που τίθεται είναι μπορούμε να βρούμε νομική βάση ώστε να έχουμε κοινή προμήθεια εμβολίων ούτως ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια που έγιναν την τελευταία φορά όπου ορισμένοι είχαν τεράστιου αριθμού πλέον στη διάθεσή τους, περισσότερα εμβόλια από όσα χρειάζονταν και άλλοι δεν είχαν. Και βεβαίω έπαιξε ένα ρόλο και η κερδοσκοπία και που παίζει ρόλο. Κάθε φορά δηλαδή που ξεσπά μια επιδημία και που οι τιμές εκτοξεύονται. Ορισμένες χώρες μέλη θυμούμε και την εμπειρία τη δική μου. Ορισμένε χώρε επλήγησαν από τις τιμές που θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν, που θα είχαν αποφύγει εάν υπήρχε αυτή η κοινή προμήθεια, που θα ήταν βεβαίως και μία δείγμα, ένα δείγμα μάλλον ε, αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών. Ευχαριστώ. Θυμήσατε πως η παραποίηση προϊόντων πλήττει ιδιαίτερα τους παραγωγούς μας ιδίως στις τιμές κρίσης. Αλλά όταν μιλάμε για παραποίηση ιδίως τροφίμων, αλλά και για ιατρικά εργαλεία, έχουμε να κάνουμε και με θέματα ασφαλείας. Παρόλα αυτά, έχουμε κανόνες. Στην Ιταλία κατασχέθησαν 24 εκατομμύρια κιλά παραποιημένων προϊόντων, που αντιστοιχούν σε 840 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αξία 840 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη δημοσιογεία στην Ευρώπη και για την ε, ασφάλεια της ιστορικής αγοράς. Κύριε Μπόργκ. Ευχαριστώ. Γνωρίζω τις ε, δυσκολίες αυτές. Δυσκολίες που δημιουργούν και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού επίσης. Διότι όσοι συμμορφώνονται με τον νόμο, ουσιαστικά αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με όσους δεν σέβονται τον νόμο. Έχουμε αυστηρότατους κανόνες ελέγχων και εκτός των χρόνων μας αυτά τα γεωργικά προϊόντα. Όμως αυτό δεν προβλέπεται για τα εισαγόμενα προϊόντα που δεν ε, εμπίπτουν στην κατηγορία των τροφίμων. Δεν θα έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένο από την υλοποίηση των κανόνων, αλλά εντυπωσιάζομαι το γεγονό ότι εκατομμύρια επί εκατομμυρίων παραποιημένα ή επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να κατασχεθούν και έχουμε καταφέρει να τα κατασχέσουμε με τη συνεργασία των αρχών. Αυτά προξενούν και οικονομικές ζημίες στις διάφορες χώρες. Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές συσκευές, γιατί τώρα δεν βρίσκω τον Ιταλικό όρο, τα ιατρικά εργαλεία, Εδώ υπάρχουν κάποια τέτοια μηχανήματα που ε, έχουν υψηλό ε, ποσοστό, ε, έχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου. Μιλάμε για την ασφάλεια του κοινού εδώ. Θα πρέπει λοιπόν οι μηχανισμοί να είναι αυστηρότεροι ακόμη από αυτούς που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Προέκυψαν κρούσματα και μάλιστα τρομακτικά προϊόντων που δεν ήταν γεωργικά, τα οποία δημιούργησαν προβλήματα σε παιδιά. Ή άλλε ιατρικέ συσκευέ που κάλεσαν θανάτου εκατοντάδων γυναικών. Ναι, ε, απαντήσατε με τρόπο ευφιέστατο. Αναφερθήκατε σε ορισμένες οδηγίες και αρκετούς κανόνες, είπατε όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους για θέματα όπως αυτό της άμπλωσης. Είπατε ότι θα σεβαστείτε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μα ο καθένας ε, θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό στο κολέγιο των επιτρόπων. Είπατε ότι το θέμα των αμβλώσεων είναι κάτι που πρέπει να το επιλύσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, όμως αφορά όλες τις γυναίκες. 70 εκατομμύρια γυναίκες χάνουν τη ζωή τους ετησίως στον κόσμο, διότι ακριβώ δεν υπάρχουν σαφείς νόμοι για τις αμπλώσεις. Δεν επιτρέπουν τις αμπλώσεις. Ε, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών σχετικά. Κύριε Μπόρκ, δύο λεπτά. Είναι θέμα ευφυΐας, αλλά όχι απλώς αν είναι κανείς ευφυής ή έξυπνος. Ε, είναι θέμα σεβασμού των ε, συνθήκων για τα θέματα αυτά. Το αν κάποιες πρακτικές επιτρέπονται ή όχι, είναι κάτι που το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Δεν έφτιαξα εγώ τις συνθήκες. Τις συνθήκες αυτές τις κυρώσαν τα κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε, δεν είμαστε ακόμη ομοσπονδία κρατών. Είμαστε μία σούι generis ε, οργάνωση κυρίαρχων κρατών που έχουν ακόμη την πλήρη κυριαρχία τους σε πολλά θέματα. Κάποιες φορές υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της κοινότητας, αλλά κάποιες φορές υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα ή όπως στην περίπτωση των υπηρεσιών υγείας, ό,τι και αν πιστεύετε εσείς, εγώ, ο καθένας, είναι ζήτημα όπου οι υπηρεσίες μου δεν μπορούν να εμπλακούν εφόσον διοριστώ επίτροπος. Δεν μπορούν να παρέμβουν στις υπηρεσίες υγείας. Άλλο για την υπηρεσία διασυνοριακής παροχής ε, υγείας που θα πρέπει να υλοποιήσουμε και άλλο ότι κάνουν τα κάτι μέλη στον δικό τους τομέα. Δηλαδή, επανειλημμένος και διαρκώς ο κάθε επίτροπος, όλοι οι επίτροποι και είδα τις κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις που έχουν τεθεί για τέτοια ευαίσθητα ηθικά ζητήματα, πάντοτε έδιναν την ίδια απάντηση. Άσχετα με την προσωπική υπεποίθηση άποψη του καθενό. Είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση σε επίπεδο κράτου μέλου. Ο καθένα από εμά έχει τι δικέ του προσωπικέ προτιμήσει. Όμω δεν μπορούμε όλοι να ε, υποχρεωθούμε να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όμω εγώ αυτό που σα λέω είναι θα σεβαστώ τι συνθήκε. Δεν θα παρέμβω σε προβλήματα που ενδεχομένω ήδη υπάρχουν, διότι θα ήταν παράνομο και δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Ευχαριστώ κύριε Φλόρεντ. Δόκτωρ Μπόρκ, τελειώνουμε σιγά σιγά. Πρώτα πρώτα επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για όλη όλα όσα μπορέσατε και απαντήσατε εδώ. Έχουμε τώρα την αρχή της ευθύνης του παραγωγού. Μπορείτε να φανταστείτε στο μέλλον ένα μέρος των δαπανών υγείας για τα προϊόντα καπνού να επιβαρύνουν τα προϊόντα καπνού. Είχαμε συνεργαστεί καλά με τον προκάτοχό σας. Γι' αυτό ρωτώ, τι υποστήριξη μπορείτε να προσφέρετε όπως ώστε να μπορέσει ο προκάτοχός σας να έχει πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που τον αφορούν για να μπορέσει να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ευχαριστώ κύριε εσείς. Για τη δεύτερη σας ερώτηση κύριε Φλόρεντς. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Διότι συμμορφώνομαι με τους νόμους του οργάνου σας και αυτοί θα ισχύσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, έρχομαι σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Εάν είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να δηλώσω τίποτε απολύτω σχετικά. Είπα ήδη από την αρχή ότι υπάρχει μια παρέτηση. Η παρέτηση σημαίνει ότι θα χρειαστεί αντικατάσταση και τα δύο θέματα, όπως είπε και ο πρόεδρός σας προηγουμένως, θα πρέπει να διακριθούν απολύτως το ένα από το άλλο. Δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο. Σας βεβαιώ κύριε Φλόρεντς ότι η θύρα μου θα είναι ανοιχτή, όχι μόνο σε εσά, σε όλους τους ευρωβουλευτές για θέματα τα οποία άπτονται του χαρτοφυλακία μου και όχι διότι αυτό είναι πολιτικά σκόπιμο για μένα, αλλά διότι είναι και το σωστό. Υπήρξα και είμαι βουλευτής επί μια εικοσαετία. Έχω συνηθίσει να υφίσταμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά είμαι και ο ίδιο βουλευτή, διότι ακολουθούμε το βρετανικό σύστημα που για να είναι κανεί υπουργό πρέπει να είναι και βουλευτή. Εμένα μου φαίνεται σωστό αυτό, γιατί σημαίνει ότι πάντοτε πρέπει κανεί να είναι σε εγρήγορση και να θέτει υπό την δοκιμασία τη εξέταση των ψηφοφόρων του τα όσα προτείνει. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδηγία που αναφέρατε, θεωρώ ότι Όλοι το αναμένουν αυτό και ως ένδειξη, ως δείγμα μάλλον αξιοπιστίας. Διότι εάν κάτι, κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει κάποιος λόγος που καθυστερεί η οδηγία θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν έχουν δίκιο. τα όργανα που συμμετέχουν στην συναπόφαση, Κομισιόν και Κοινοβούλιο, δεν προτίθεται να αποδυναμώσουν την οδηγία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην pipeline. Dagmar Δύο θέματα για την υγεία των ζώων. Συμφωνείτε ότι η φυστάμενη νομοθεσία όπως αυτή για τα καλλιντικά πρέπει να εφαρμόζεται και να εφαρμοστεί χωρίς αλλαγές. Και το τελευταίο τμήμα της να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον επόμενο Μάρτιο. Δεύτερο, μεταφορά ζώων μας έχουν διαβεβαιώσει δύο από τους προκατόχους σας ότι θα επενεξεταστεί ο χρόνος μεταφοράς των ζώων και έχουμε και νομοθετική πρόταση και πέραν των όσων αναφέρατε προηγουμένως. Θα υποβάλλετε πρόταση για τη μεταφορά ζώων. Ευχαριστώ. Ο συνήθως σύντομη και περιεκτική. Ευχαριστώ κύριε Ρότ. Κύριε Ρότ Μπέρντ. Για το πρώτο θέμα. Πρώτον, ευημερία ζώων και νομοθεσία περί καλλιντικών. Είπα ότι η διαδικασία είναι τόσο δυσκίνητη. Να περάσει δηλαδή η νομοθεσία από όλη αυτή τη διαδικασία. Βεβαίω υπάρχει και ένα λόγο. Διότι είναι ένα νόμο που θα εφαρμοστεί μοναχά στη Γερμανία ή στη Μάλτα. Θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα είναι λογικό να είναι μακρά και επίπονη η διαδικασία. Και όταν γίνει, ε, εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή και με κάποιε μεταβατικέ περιόδου, προσπαθούμε καμιά φορά να επινοήσουμε κάτι για να αποφύγουμε την εφαρμογή. Εγώ βρίσκω ότι αυτό δεν είναι έντιμο. Φάκτα λέξ inventa fraus. Δηλαδή από τη στιγμή που ισχύει ένα νόμο, προκαλεί και μια τάση επινόησης απατών. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Νομίζω ότι η απαγόρευση πρέπει να εφαρμοστεί όπως έχουν αποφασίσει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις συνέπειες της απαγορεύσεως διότι το λεγόμενο impact assessment πρέπει να λειτουργεί και μετά την εφαρμογή. Και υπάρχει ένας άλλος λόγος. Εάν δεν το πράξουμε, η βιομηχανία δεν θα προσπαθήσει ποτέ να βρει εναλλακτικά μέσα δοκιμασίας εκτός των πειραματοζώων. Στα αγγλικά, γιατί δεν είμαι Άγγλος εγώ βέβαια, στα αγγλικά λέμε ότι η ανάγκη είναι η μάνα της επινοητικότητας. Όταν είσαι υποχρεωμένος να επινοήσει κάτι άλλο, θα πάρει χρόνο, αλλά θα το επινοήσει τελικά. Άρα λοιπόν, ναι, η απαγόρευση πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2013. Τώρα, για την μεταφορά ζώων. γνωρίζω ότι οι υποσχέσεις επανέρχονται και σε κυνηγούν ως μπούμεραγκ. Δεν θέλω λοιπόν να έρθετε και να μου πείτε «Α, υποσχέθηκες». Θα δω πάντως τι μπορούμε να κάνουμε μαζί με άλλους επιτρόπους και σχετικά με την μελέτη επιπτώσεων για την βελτίωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων. Δεν δεσμεύομαι για τις 8 ώρες, θα προσπαθήσω ωστόσο με κάθε τρόπο να βελτιώσω την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος, αλοχιάσκατος ο Μίχαλ Ζέβερ. Μάλιστα, είμαι τελευταίο. Επιτρέψτε μου να πω ότι παρακολούθησα μια πολύ ισχυρή performance. Όχι μόνο FE, αλλά αποδείξατε ότι θα όντω μπορούμε να σε πιστέψουμε δηλαδή ότι θα λειτουργήσετε στη βάση των συνθήκων και του χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Μακάρι να σας είχαμε ε, ε, Υπουργό Περιβάλλοντος στη χώρα μου. Εμεί βεβαίω είμαστε αρμόδιοι εδώ ως Επιτροπή και για περιβάλλον και για υγεία. Θα υποστηρίξετε λοιπόν τα αιτήματά μα. Δεύτερο, πώ θα διαμορφώσετε τι σχέσει συγκεκριμένα με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή περιβάλλοντο. Θα διαβουλεύεστε μαζί μα πριν να καταθέσετε προτάσει και πόσο συχνά θα μα επισκέπτεστε, πόσο εντατικέ σχεδιάζεται να είναι οι επαφέ μαζί μα. Για μα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το Κοινοβούλιο ότι ακούτε τις αιτήσει μας, τα αιτήματά μας δηλαδή, γνωρίζουμε ότι εμείς στο θεσμικό πλαίσιο δεν έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας, αλλά πώς θα συνεργαστείτε μαζί μας. Ευχαριστώ και Ζέμπερ. Πολλές ερωτήσεις βέβαια, πυκνές. Δύο λεπτά, ο υποψήφιος επίτροπος. Υποψήφιος επίτροπος, διορθώνω λέει πρόεδρος γιατί είπε επίτροπος. Βεβαίως, ουδής λογικός άνθρωπος θα έλεγε όχι δεν θα έρχομαι να διαβουλεύω μαζί σας. Αλλά θα πρέπει επίσης να είμαι έντιμος απέναντί σας. Θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μου όσο μπορώ καλύτερα για να διατηρήσω τον σύνδεσμο αυτό με το μόνο πραγματικά δημοκρατικό και άμεσα εκλεγμένο όργανο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκλεγμένο από τους λαούς και που βεβαίως έχει δει να αυξάνονται οι αρμοδιότητες του στην διαδικασία συναπόφαση μετά από την θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Ωστόσο, θα ήθελα να πείσω τον καθένα και την καθεμιά από εσά και εσά που συμφωνείτε και εσά που δεν συμφωνείτε μαζί μου. Όσοι θα είστε υπέρ τη εγκρίσεώ μου και όσοι θα διστάσετε. Θα σα πω ότι αισθάνομαι άνετα στο κοινοβουλίο, διότι είμαι ο ίδιο κοινοβουλευτικό. Δεν λέω ότι οι επίτροποι οι οποίοι δεν πήγαν να χτυπήσουν τις πόρτες των εκλογέων τους δεν είναι άνθρωποι κανεί να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Θα έλεγα ότι ο γυναικολόγος δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει να γεννά μια γυναίκα διότι ο ίδιος δεν μπορεί να έχει γεννήσει ποτέ. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είμαι υπόλογος απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ότι με ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Αυτό σας προσφέρει ένα πλεονέκτημα. Πρέπει να το εκμεταλλευτείτε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Αν το αφήσετε να αποθάνει βεβαίως δεν θα υπάρχει διαφορά. Αλλά αν όμως πραγματικά αισθάνεστε ότι είστε κοινοβουλευτικός που σας έχει εκλέξει ο κόσμος για να εκπληρώσετε ένα σκοπό, έτσι θεωρώ εγώ, τότε αυτό επιφέρει κάποια διαφορά στις σχέσεις κάποιου προσώπου με ένα κοινοβούλιο. Εγώ λέω πάντα στους συνεργάτες μου, μα μην διαμαρτύρεστε όταν λαμβάνουμε κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις, διότι οι ερωτήσεις επισημαίνουν τις αδυναμίες του Υπουργείου. Και ε, ελπίζω ότι τα λόγια αυτά θα μπορέσουν να μεταμορφωθούν και σε πράξη, αλλά βέβαια αυτό θα το αποφασίσετε εσείς πλέον αργότερα, εφόσον με εγκρίνετε, εάν δηλαδή τήρησα τι υποσχέσεις μου. Ευχαριστώ κύριε Μπόρκ. Έχουμε φτάσει στο τέλος φτάσει στο τέλος των γύρων ερωτήσεων. Θα λάβετε τώρα το λόγο για πέντε λεπτά. Μπορείτε να περιοριστείτε και σε λιγότερα λεπτά αν θέλετε. Για μια τελική δήλωση. Μετά θα λάβει το λόγο ο κύριος Χάρμπορ και μετά θα μιλήσω. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ αυτή την ημέρα που είναι μέρα αφιερωμένη στην Ευγένεια που ήσασταν κι εσείς απέναντί μου τόσο καλή. Το θέμα δεν είναι να είναι κανείς ε, ευφύης, ξύπνιος. Εγώ προσπάθησα να είμαι ο μου. Και πρέπει να σας πω και πιστέψτε με ότι αυτό που βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει καμία κρυφή ατζέντα. Τίποτα κρυφό δεν υπάρχει. Προσπάθησα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας όσο γίνεται με περισσότερη πληρότητα. Συγγνώμη για τα όποια λάθη. Συγγνώμη αν δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά βέβαια μέσα σε τρεις εβδομάδες υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να μάθει κανείς. Πάντως, Κατάλαβα το πνεύμα πίσω από τις ερωτήσεις σας που είχα να κάνω με το χαρτοφυλάκιό μου. Δεν είναι θέμα εξωτερικών υποθέσεων, είναι μια απτή πραγματικότητα. Οι κοινοβουλευτικοί παντού ανά τον κόσμο, εφόσον φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους, έχουν πάντα μια ανοιχτή ε, γραμμή με τους πολίτες. Όταν ε, υποβάλλουμε μια πρόταση, πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο και στην βιομηχανία. Και συμφωνώ με το σχόλιο που έγινε. Εφόσον ε, με εγκρίνεται, και μου δώσετε την χαρά να σας υπηρετήσω, θα θυμάμαι πάντα την παρατήρηση αυτή, ότι όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει κάτι, έχει και τη δημοκρατική σφραγίδα εκατομμυρίων πολιτών και λαμβάνει υπόψη και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν ε, καθαρά και μόνο με το Κοινοβούλιο. Η δικιά μου φιλοδοξία, εφόσον με εγκρίνεται, είναι να υποβάλω μια φιλόδοξη πρόταση για τα καπνά, πρώτον, και δεύτερον, να σεβαστώ την προθεσμία του 2013 για τα πειράματα ε, στα ζώα για τα καλλιτικά, τρίτον κλωνοποίηση για τα μέσα 2013 που έχει άμεση σχέση με τα θέματα προστασίας των ζών και τέταρτον, και αυτό θα είναι το πιο δύσκολο, θέλω να επενδύσω περισσότερο στο θέμα της ε, εφαρμογής των ε, κανόνων. Ελπίζω να σας έδειξα ότι από την αρχή της καριέρας μου στην ε, Μάλτα ήμουν 17 όταν έγινα μέλος στο κόμμα, πάντα υποστήριζα και προωθούσα τις ευρωπαϊκές ιδέες και σε εύκολους καιρούς και σε δύσκολους καιρούς. Και αναλαμβάνω την υποχρέωση να προωθήσω τις ευρωπαϊκές αξίες και αυτές της μη διάκρισης. Είμαι έτοιμος και βασίζομαι σε στενή συνεργασία μαζί με εσάς στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι που με υποδεχτήκατε τόσο καλά και προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας στο μέλλον. Thank you very much. Ο πρόεδρος Γκρότε. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου Μάλκον Χάρμπορ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρώτα, επιθυμώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος και σας ως Πρόεδρο που επιτρέψατε μέλη της δικής μου Επιτροπής να παίξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, στοχευμένο ρόλο στην ακρόαση. Εμείς λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα των καταναλωτών. Επανέρχομαι λίγο σε κάτι που είπε ο κ. Μπόρκ στην αρχή της ομιλίας του, όταν είπε ότι το χαρτοφυλάκιό του είναι Europe on the ground, Νομίζω προσεγγιστήκαμε πολύ. Μας δώσατε πολύ τροφή για σκέψη για τις ε, συνεδριάσεις μας. Αναλάβατε και πολλές σημαντικές δεσμεύσεις απέναντί μας. Και εφόσον εγκριθεί ο διορισμός σας, θα επανέλθουμε. Και οι συζητήσεις που όπως υποσχεθήκατε θα κάνετε με το Συμβουλίο θα επανέλθουν και στα θέματα αυτά. Εφόσον το Κοινοβούλιο βέβαια το εγκρίνει. Και για σας, Πρόεδρε Γκρότε, συγχαρητήρια για την πολύ καλά οργανωμένη ακρόαση που επέτρεψε να εξετάσουμε πολλά και ποικίλα θέματα, όχι μόνο αυστηρά της δικής σας Επιτροπής, αλλά και άλλων επιτροπών και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Μια διοικητική τώρα ανακοίνωση. Προσκαλώ όλους τους συντονιστές της Επιτροπής ενία Αγοράς να συναντηθούν μαζί μου στις 6 και 4 στην αίθουσα 6Q2, όπου θα αναλύσουμε την ακρόαση μεταξύ μας και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε και με τους ε, ε, συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 7. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Ο πρόεδρος Κρότε, ευχαριστώ αγαπητέ Μάλκολμ. Τελειώνοντας επιθυμώ να πω ότι ήταν μια ημέρα επιτυχημένη, ότι εδώ σήμερα αποδώσατε πραγματικά εξαιρετική performance και εν ώψη της συντομίας του χρόνου σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προετοιμασίας σας, που ήταν λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Νομίζω πράγματι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Δείξατε ότι διαθέτετε τεχνικές γνώσεις, αλλά και προσωπικές ικανότητες. Το, καθαρίσατε, το ξεκαθαρίσατε αυτό σήμερα Και σε ό,τι αφορά την περίπτωση Τζον Ντάλι, με τον οποίο καλά συνεργαστήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου προσήλθε πάντοτε και όπου έχερε μεγάλη εκτιμήσεω, καλώ κάναμε και διακρίναμε τι δύο αυτέ περιπτώσει. Όπω ζητήσατε και, και ορισμένοι εξημών, να του προσφερθεί δίκαιη πρόσβαση στα έγγραφα. Σήμερα συζητήσατε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό για μας να έρθει στο τραπέζι μας η οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Αναλάβατε δεσμεύσεις και για άλλα πράγματα. Θα σας μετρήσουμε σε σύγκριση με αυτές τις δεσμεύσεις σας. Δεν θα έχουμε προκαταλήψεις. Όπως είπα θα δούμε τι θα κάνετε. Θα είστε ο Επίτροπος όλων των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρώπης. Και το ύψιστο αγαθό που διαθέτουν οι άνθρωποι αυτοί είναι η υγεία τους. Και γι' αυτό ο τομέας αυτός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος. Αναλαμβάνεται μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι εγκαρδίως για την έντιμη ακρόαση που μπορέσαμε να διεξαγάγουμε σήμερα, την ε, ευγένεια που ίσχυσε ε, σήμερα, όπως ε, εξήγησε προηγουμένως ο κύριο Παρνιό, το πρωί μάλλον, Ευχαριστώ συνολικά 15 υπηρεσίες οι οποίες στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους μπόρεσαν να οργανώσουν μια ακρόαση η οποία έρεται στο ύψος των περιστάσεων. Για τους συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος ανακοινώνω ότι θα συναντηθούμε στις 7 εδώ στην παρούσα αίθουσα 2Q2 για να κάνουμε την αξιολόγηση της ακροάσεως. Σας εύχομαι σε όλες και όλους οι οποίοι έχετε τελειώσει την εργασία σας. Καλό βράδυ.